Good gentlemen. May I ask you... Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Κυρίζω την έναρξη της απογευματινής συνεδρίας της Επιτροπής ε, της Επιτροπή μας, ε, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διαταξή μας είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Γιάκ Αμπ, Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης, ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις προτεραιότητες της Θονικής Προεδρίας. Δεν θα μιλήσω περισσότερο για την Εστονική Προεδρία, γιατί θα μας ε, πει ε, σχετικά ο ε, Υπουργός. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω τα διαδικαστικά. Θα δώσουμε το λόγο στον Υπουργό για την παρουσίασή του. Στη συνέχεια θα, δοθούν, θα δοθεί ο λόγος στα μέλη της Επιτροπής να ξεκινούμε με τους συντονιστές. Θα θέσουν τα ερωτήματά τους και εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και σας παρουσιάζω τις προτεραιότητες της πρώτης εσθονικής προεδρίας ε, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να ξεκινήσω με τις γενικές ε, προτεραιότητες της Προεδρίας και στη συνέχεια να περάσω σε θέματα που είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικά για την Επιτροπή σας. Τα κύρια θέματα της Προεδρίας μας ε, συνάδουν ε, με τον οδικό χάρτη της Πρατισλάβας ε, και η, δουλειά μας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα έχει ως γνώμονα τέσσερις βασικές αρχές. Η πρώτη προτεραιότητα για την Εστονία κατά την Προεδρία της είναι μια ανοιχτή και καινοτόμως ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περισσότερο από μία οικονομία, αλλά μία ισχυρή και καινοτόμως οικονομία μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια, την ειρήνη ε, την ε, σταθερότητα και την ευημερία. Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που απαρτίζεται από 500 εκατομμύρια καταναλωτές είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας. Ε, είναι ένας θεμέλιος λίθος της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι επιχειρήσεις μας μπορούν να ανθίσουν μόνο σε ένα απλό, προβλέψιμο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί πολύ συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τομέα αυτό. Η δεύτερη προτεραιότητα της Προεδρίας μας είναι η ασφάλεια ε, της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε πάνω, εδώ και πάνω από 60 χρόνια ως ε, ε, ένα εγχείρημα υπέρ της ειρήνης και τα ζητήματα ασφάλειας εξακολουθούν να είναι τμήμα των ε, προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν και τα σχετικά προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταναστευτική κρίση και για να μπορέσουμε να είμαστε επιτυχείς πρέπει να συνεργαστούμε. Ένα ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης είναι προς όφελος όλων μας. Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ασφαλή και να την κάνουν καλής διαχείρισης για να μπορούμε να είμαστε ασφαλείς αλλά να υπάρχει και ελευθερία κυκλοφορίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η ποιότητα των ε, συστημάτων πληροφόρησής μας είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία ε, ως προς αυτό. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, η τρίτη προτεραιότητα της Εστονικής Προεδρίας είναι η ψηφιακή Ευρώπη και η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων. Έχουμε ένα διεξοδικό ψηφιακό πρόγραμμα που είναι ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ε, εσφωνικό, αν θέλετε, στην Προεδρία μας. Για μας είναι ένα ζήτημα εγκάρσιο, το οποίο είναι σημαντικό για κάθε τομέα. Το επίκεντρο του ψηφιακού προγράμματός μας είναι το πακέτο ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η ψηφιακή ανάπτυξη συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, μας δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουμε διασυνοριακές συνεργασίες και το, ε, συγγνώμη, συναλλαγές και ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, θέλουμε υπό ένα ψηφιακό πρίσμα να δούμε ό,τι κάνουμε στο πλαίσιο της Εστονικής Προεδρίας μας. Οι ψηφιακές λύσεις μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι καλύτερο και ευφιέστερο σε κάθε τομέα. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω την τέταρτη προτεραιότητά μας. Η τέταρτη και τελική τελευταία προτεραιότητα είναι μία χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας, αλλά μία αηφόρος και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη ε, είναι, όπως και το ψηφιακό κομμάτι, ένα εγκάρσιο θέμα, ίσες ευκαιρίες και ένα ισότιμο περιβάλλον διαβίωσης είναι ε, κάτι που είναι προς όφελος όλων των ε, ε, πολιτών. Ελπίζω να κατάφερα να σας κάνω μία μικρή σύνοψη των βασικών ε, στοιχείων ε, του προγράμματος της Προεδρίας μας. υποθέτω βεβαίως ότι εσείς μπορεί να με ρωτήσετε σε αυτό το σημείο και τι έχετε να πείτε για την ε, Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Πρέπει να μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα διατομεακό θέμα το οποίο συνεισφέρει υπέρ πολλών ευρωπαϊκών στόχων. Η πολιτική συνοχή είναι καταρχάς, έχει καταρχάς στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες και στις περιφέρειες και στη μείωση των διαφορών των επιπέδων ανάπτυξης, παράλληλα συνδέεται με την αηφόρο ανάπτυξη και τις ίσες ευκαιρίες. Μεταξύ άλλων, η πολιτική ε, συνοχής ε, συμβάλλει και στην προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας. Η ψηφιοποίηση και η χρήση ηλεκτρονικών λύσεων ε, μας έχουν βοηθήσει να εφαρμόσουμε την περιφερειακή πολιτική καλύτερα και να αυξήσουμε την ορατότητά της. Όπως βλέπετε, η πολιτική συνοχή συνδέεται με πολλές από τις προτεραιότητές μας. Η πολιτική συνοχή ε, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εστονικής οικονομίας και επίσης ε, στην ε, διεξαγωγή διαρθρωτικών ε, αλλαγών. Η πολιτική συνοχής ε, μας βοήθησε στην ανάκαμψη της, ε, από τη σοβαρή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και πιστεύω ότι η Εστονία είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς η πολιτική συνοχής από κοινού με μία στέρεα οικονομική πολιτική μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική σύγκληση. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Έχουμε και δύο ευρύτερε προτεραιότητε στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή. Πρώτον, θα θέλαμε να συνεχίσουμε τις συζητήσει ε, περί απλούστευσης, αποτελεσματικότητας και μέλλοντος της ε, πολιτικής ε, συνοχής. Η Προεδρία μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής η Προεδρία μας έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα προς το μέλλον. Οι προηγούμενες Προεδρίες έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για το μέλλον. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς βεβαίως το σκέφτεστε, το γνωρίζουμε και είμαστε ανοιχτοί στις ιδέες σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει έγγραφα συζήτησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εξή έγγραφα, όπως για παράδειγμα πολύ ε, ε, ανακοινώσεις όσον αφορά ε, την ψηφιοποίηση στις άκρος απομακρυσμένες περιοχές, όπως επίσης και η έβδομη έκθεση συνοχής. Η συνοχή πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειών της, αλλά παράλληλα πρέπει να είναι και κοντά στους πολίτες είναι μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο, όμως ο αντίκτυπος είναι πανευρωπαϊκός. Στο μέλλον, η αποτελεσματική πολιτική συνοχής πρέπει να έχει σαφείς στόχους, λογικούς και διαφανείς κανόνες και δεν θα έπρεπε να υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία. Αυτή είναι η πολιτική συνοχής ε, για την οποία αγωνιζόμαστε. Αυτή είναι η πολιτική συνοχής που είναι απαραίτητη για τους πολίτες μας και σημαντική για αυτούς. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εχθές η σύσταση της ομάδας υψηλού επίπεδου για την απλούστευση δημοσιεύθηκε. Περιμέναμε αυτήν ε, την δημοσίευση, γιατί η απλούστευση είναι ένας τομέας ε, που επιδέχεται ε, βελτιώσεων ε, είναι, ένα, ένα, είναι κοινό το όφελος από αυτήν ε, και πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό οι συζητήσεις για την πολιτική συνοχής να λάβουν χώρα σε ένα πιο επίσημο επίπεδο. Θέλουμε να συζητήσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχής το Νοέμβριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα ε, αφορά ειδικότερα την πολιτική συνοχής ε, και μάλιστα αυτό θα είναι και το θέμα του ε, Συμβουλίου αυτού. Η πολιτική συνοχής μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε την εφαρμογή της και την εξέλιξή της ως τώρα και να την αναθεωρήσουμε έχοντας στο μυαλό μας ένα σαφές όραμα θα έχουμε λιγότερο επίσημες συζητήσεις Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Θα γίνουν ε, συναντήσεις για τις οδηγίες ε, εδαφικής πολιτικής, πολιτικής συνοχής ε, και εδαφικής ανάπτυξης. Ε, θα γίνει πρώτη αναθεώρηση του προγράμματος αστικής ανάπτυξης για τις αρχές του επόμενου έτους. Ο κανονισμός Omnibus έχει ήδη συζητηθεί αυτός από εσά και έχει, έχετε υποβάλει και την άποψή σας. Χάρη στη δουλειά της Προεδρίας της Μάλκας έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο στη διαδικασία διαδικασία αυτή, στο οποίο μπορούμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι αρχές της Προεδρίας μα ήδη. Πρέπει να πω ότι είναι μια διεξοδική πρωτοβουλία. Κατά την άποψή μου, ε, η απλούστευση που προτείνεται από την πρωτοβουλία είναι προς όφελος όλων. Αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. η αντίδραση στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι πολύ ενθαρρυντικό όταν σκέφτεται κανείς το μέλλον. Εμείς μέσω στη συνεργασία μας θεωρούμε ότι θα υπάρξει ταχεία πρόοδος. Οι αλλαγές έχουν γίνει πολύ που έχουν γίνει πολύ σημαντικές για τους δικαιούχους και καθιστούν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ευκολότερη και πιο ευέλικτη. Εκτός από αυτές τις δύο προτεραιότητες, θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαστε, παραμένουμε δεσμευμένοι ε, σε χρηματοδότηση από τα ε, ταμεία ε, αλληλεγγύης για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω του σεισμού στην Ιταλία και ελπίζουμε ότι θα επισπευθούν οι σχετικές συζητήσεις στο Συμβούλιο. Επίσης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ενημερώνουμε τους πολίτες μας για τα επιτεύγματα της πολιτικής με πολύ χαρά μπορώ να σας πω σήμερα ότι πάνω από το 80% των Εστονών γνωρίζουν την υποστήριξη που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Εστονία και η πλειοψηφία ε, αυτών ε, πιστεύουν ότι αυτό έχει μια θετική έχει θετικό αντίκτυπο στην Εστονία και στην οικονομική μας ανάπτυξη. Αυτά είναι εξαιρετικά αποτελέσματα. όλοι οι επιβάτες που έρχονται μέσω του αεροδρομίου του Ταλίν στην Εστονία μπορούν να δουν και μία έκθεση για τα επιτεύγματα της ε, πολιτικής συνοχής. Ελπίζουμε ότι θα την απολαύσετε αυτήν την έκθεση κατά την επίσκεψή σας στο Ταλίν αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πολιτική συνολή, συνοχής που εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές αξίες, ε, που είναι αποτελεσματική, και έχει προστιθέμενη αξία, είναι πολύ σημαντική για όλους μας και εμείς θεωρούμε εξαιρετικά πολύτιμη τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο αεροδρόμιο του Ταλίν την έκθεση. Θα ήθελα τώρα να αρχίσουμε τη συζήτηση. Ε, με τους συντονιστές, θα θέσουν τις ερωτήσεις και θα κάνουν τις συστάσεις τους. Κύριος Βανίστελο κύριος Βανίστελο ο πρώτος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα την εισαγωγή σας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ε, είδα και τους ε, στόχους σας οι οποίοι νομίζω ότι ταιριάζουν πολύ καλά με την εικόνα που έχουμε για τη χώρα σας. Επομένως, ε, ήταν ικανοποιητικό να διαβάσω και το κείμενο για το πρόγραμμά σας. Θα μπορούσα ίσως να σας διαβάσω και κάποια πράγματα ε, για τη συνοχή που αναφέρεται εκεί. Υπάρχουν πολύ καλές ιδέες. Λέτε ότι χρειαζόμαστε συζήτηση για τη συνοχή στα αγγλικά λέτε λαμβάνοντας υπόψη την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τους λόγους για τους οποίους ε, ε, υποστηρίζουμε ε, μια ισχυρή πολιτική συνοχής. Πρόκειται για σαφή διατύπωση, η οποία εκφράζει σαφέστατα την θέση σας και εμείς τα υποστηρίζουμε αυτά. Ε, κοιτώντας όμως λίγο πιο προσεκτικά το κείμενο, θα ήθελα να συμφωνήσω με την ε, πρόεδρο ε, για την ε, πρόσκληση στο Ταλίν, αλλά η ουσία που είναι στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων σας. Στην προηγούμενη Προεδρία, στη Μαλτέσκη Προεδρία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε στενά στις συζητή, ενεργά στις συζητήσεις και είχαμε και μια αρκετά αισιόδοξη συζήτηση για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε και κάποια βήματα περαιτέρω. Αναφέρεστε στην απλοποίηση. Και είστε και υπεύθυνοι για το Omnibus, το οποίο περιλαμβάνει και αυτό μία σειρά από προτάσεις πολιτικής ε, στον τομέα αυτό και η πρόταση είναι να μπορέσετε να τα ολοκληρώσετε αυτά ε, αρκετά σύντομα στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ε, ε, από πλευράς πολιτικής θα έχουμε την 7η έκθεση συνοχής και η ερώτησή μου είναι πώς μπορείτε να μας εξασφαλίσετε ότι θα συμμετέχουμε κι εμείς ε, αναφέρεται ένα άτυπο Συμβούλιο Υπουργών και αυτό είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να περιμένουμε για ένα τέτοιο έγγραφο. Δεν ε, έχω δει κάτι εδώ, δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί κάπου σε αυτό αλλού. Ε, θα μπορούσατε να μας ε, κάνετε κάποιες συγκεκριμένες προσκλήσεις, ώστε τα, οι μέλη της Επιτροπής και η Πρόεδρος να μπορέσουν να συνεισφέρουν ε, στην ε, συνεδρία των Υπουργών στο Συμβούλιο και θεωρώ ότι αυτή η προετοιμασία θα μπορούσε ε, να μας βοηθήσει να σας υποστηρίξουμε. Είναι καλό να υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ μας, αλλά χρειάζεται και να κάνει και αυτό, ο καθένας αυτό που του αναλογεί. Αναφερθήκατε επίσης στο ψηφιακό θεματολόγιο. Πρόκειται για κάτι το οποίο ενδιαφέρε πάντα το Κοινοβούλιο. Είχαμε και το Connecting Europe Facility η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει τότε 10 δις ευρώ ε, όταν ήταν επίτροπος η Νέλη Κρούς για το θέμα αυτό. Και το Συμβούλιο το διέγραψε αυτό, ενώ εμείς ως Κοινοβούλιο είχαμε βάλει τα θέματα τεχνολογίας της πληροφορικής και της κοινωνίας και το ψηφιακό ε, θεματολόγιο ε, στη δεύτερη θέση στις προτεραιότητές μας. Το Κοινοβούλιο λοιπόν ε, έκανε αυτό που το αναλαγούσε, αλλά το Συμβούλιο δεν ακολούθησε. Εάν λοιπόν θέλουμε να επιτύχουμε κάποιους στόχους, πρέπει να, να, να συνεργαστούμε. Κυρία Βέστφαλ, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να σας πω, δεν είμαι συντονίστρια, αλλά πρέπει να σας πω ότι νιώθω... Ε, ότι επιβεβαιώνω αυτά που πιστεύω. Όπως ξέρετε, πριν από κάποιο καιρό ε, ψηφίσαμε για μια έκθεση ε, σχετικά με την πολιτική συνοχή. Ε, με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε η έκθεση αυτή από το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ερωτήματα. Και εσείς ήδη αρκετά είπατε για την πολιτική συνοχής. Για μας όμως υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες που είναι πολύ σημαντικές. Η απλούστευση, το είπατε κι εσείς, ε, είναι πολύ σημαντική. Εχθές ε, η ομάδα υψηλού επίπεδου παρουσίασε την έκθεσή της. Πολύ ωραία το ότι όλα αυτά που είναι σημαντικά για μας ε, και κυρίως είναι σημαντικά και για τους πολίτες, πολύ ωραία το ότι είχε απήχηση η έκθεση αυτή. Για μας όμως έχει μεγάλη σημασία και φοβόμαστε ότι δεν θα λάβει χώρα το ότι και στο μέλλον ε, θα πρέπει να στηρίζονται όλες οι περιφέρειες, όχι μόνο οι φτωχότερες και οι πιο αδύναμες, αλλά και εκείνες που αυτή τη στιγμή τα πάνε καλά, που ε, είναι καλές περιοχές, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Και αυτό ε, το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από μένα, λόγω της χώρας σας, Υπάρχουν καταστάσεις, μπορεί να εμφανιστούν καταστάσεις που απαιτούν να υπάρχει ευελιξία στα προγράμματα. Και αυτό λοιπόν εμείς το πήξαμε στην έκθεση πρωτοβουλίας. Όσον αφορά τώρα την ψηφιοποίηση, τη γενικότερη, είπατε κάτι που και εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή να υπάρχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια προσαρμογή. Αν είμαι σωστά ενημερωμένη, ε, εσείς ε, χρησιμοποιείτε ευρέω την ψηφιοποίηση, ε, σε άλλες χώρες δεν είναι αυτονόητο. Και το τελευταίο, πιστεύω, είναι το εξής. Ως κοινοβούλιο συστήσαμε μια έκθεση πρωτοβουλίας και νομίζω ότι το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης είναι καλό. Τώρα λοιπόν αυτό που παίζει ρόλο είναι να σφυριλατήσουμε ένα μέτωπο έτσι ώστε η πολιτική συνοχή στο μέλλον ε, να έχει απήχηση. Γιατί τη τελική ανάλυση αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι ε, μπορεί κανείς να λέει μόνο καλά πράγματα για την Ευρώπη, αλλά επιτόπου κρίνονται τα πράγματα. Ε, όταν οι άνθρωποι δηλαδή οι ίδιοι νιώθουν στο πετσί τους τι σημαίνει Ευρώπη. Επόμενος ομιλητής, ε, ο κύριος Βαν Μίλτενμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χτες ε, είχα ήδη την ε, χαρά να σας ε, γνωρίσω και να έχω μια πρώτη συζήτηση μαζί σας. Και πάνω σε αυτό θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή του αστικού θεματολογίου. Και τώρα έχω έτσι μια γενική εικόνα για το τι ακριβώς ε, ε, επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Νοέμβρη. Θα υπάρχει έκθεση πρόοδου για, την αστική, για το αστικό αυτό θεματολόγιο. Ε, μεταξύ άλλων έχουν δηλώσει και η Εστονία ότι ενδιαφέρονται. Εσείς θα το συμπεριλάβετε αυτό ε, όταν θα υπάρξει συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Δηλαδή προτίθεστε να το θίξω θέμα στην στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και ανεξάρτητα από το μέλλον της ε, πολιτικής ε, συνοχής ε, πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται και στη δική μας τη χώρα με την πολιτική συνοχής. Παραδείγματο χάρη τι χρειάζεστε, την πολιτική συνοχή για να εφαρμόσετε το ψηφιακό θεματολόγιο. Τι μπορεί να μάθει η Ευρώπη από εσάς ε, κατά τη διάρκεια της ε, σας. Η πρόταση για το πρόγραμμα Omnibus ε, νομίζω πολύ σωστά επισημάνατε και θέλω να κάνω έκκληση σε εσά να προχωρήσετε χωρίς καθυστερήσει γιατί η Ευρώπη ε, περιμένει να πλουστευτούν τα πράγματα και να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ λοιπόν εκφράζω την επιθυμία αυτό το θέμα να το κλείσετε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας σας. Και τέλος, ε, μια πολιτικά ευαίσθητη συζήτηση, όπου μπορώ να φανταστώ ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε, είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο Συμβούλιο, πρόκειται για την αιρεσιμότητα. Ε, έχουμε την οικονομική αιρεσιμότητα, αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αιρεσιμότητα όταν πρόκειται για το προσφυγικό. Ε, το θεωρώ σημαντικό αυτό. Στην πρόταση για το πρόγραμμα Omnibus η Κομισιόν προτείνει εκτός από την μέρημνα για τους πρόσφυγες να υπάρχει και μία ε, ζώνη ε, επενδύσεων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εσείς ε, πώς το βλέπετε αυτό και ίσως θα ήταν καλό το θέμα να τεθεί κατά τη διάρκεια της δικής σας της Προεδρίας. Ίσως να είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει ίσως παρόλα αυτά να γίνει η συζήτηση. Και τέλος ε, θέλω να ε, σας ευχηθώ καλή επιτυχία. η φιλελεύθεροι και εγώ σας εμπιστευόμαστε. Στο ονόματος της ΓΟΥ, ο κύριος Ομαρζέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κύριε Υπουργέ ε, εδώ για αυτή την ανταλλαγή απόψε στην αρχή της Προεδρίας, η οποία πρέπει να πούμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη, δεδομένων και των προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τα υπενθυμίσατε κι εσείς. Έχουμε τη μεταναστευτική κρίση, έχουμε το Brexit, έχουμε τα προβλήματα της έλλειψης ασφάλειας. Ε, δεν χρειάζεται να επανέλθω τώρα σε όλα αυτά. Οι μεγάλοι ελιγμοί ξεκίνησαν και μάλιστα ξεκίνησαν για όλες τις ε, κοινοτικές πολιτικές, ε, τις οποίες επανεξετάζουμε αυτή τη στιγμή και ξεκίνησαν και για το μέλλον, ε, για το μελλοντικό πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε πέντε εναλλακτικέ λύσεις. Για αυτά τα πέντε σενάρια, τα τέσσερα μου φαίνεται ότι δεν είναι υπέρ της πολιτικής συνοχής και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας την ε, αίσθηση για το θέμα. Ε, σας δημιουργεί ερωτηματικά, σας ανησυχεί το όλο θέμα. Ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρκετοί ανησυχούμε για το μέλλον της ε, περιφερειακής πολιτικής. Και όχι μόνον όσον αφορά τα θέματα του προϋπολογισμού, αλλά και όσον αφορά τη ε, σημασία και την έννοια που θα προσδώσουμε στη μελλοντική περιφερειακή πολιτική. Για να το πω με δύο λόγια, θέλουμε να διατηρήσουμε μία φιλόδοξη περιφερειακή πολιτική σε επίπεδο προπολογισμού, αλλά ταυτόχρονα και μία πολιτική η οποία δεν ε, θα ε, χάσει την κάθε ουσία της και πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές προτάσεις που κυκλοφορούν ε, οι οποίες θέλουν ακριβώς αυτό να χάσει την ουσία της η ε, περιφερειακή πολιτική. Θα ήθελα να ξέρω και τη θέση σας, για παράδειγμα, για την πρόταση που κυκλοφορεί ε, να διαγράψουμε τις κατηγορίες των περιφερειών. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω και τι πιστεύετε ε, όταν χρησιμοποίησαμε ε, το μαστίγιο της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, τώρα χρησιμοποιούμε το καρότο, το δέλεαρ, με προτάσεις για τις περιφέρειες οι οποίες θα σεβαστούν τα κριτήρια. Για μας αυτό ε, ουσιαστικά μας οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα και ε, για λόγους αρχής ε, αρνούμαστε κατηγορηματικά αυτή τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα η οποία εκφύσεως ε, ε, δεν συνάδει με την πολιτική συνοχής. Δεν θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχής είναι, υπάρχει για να την εντάξουμε στις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, θα ήθελα να σας σχολιάσω και λίγο το ψηφιακό θεματολόγιο και κάποια πράγματα που είπατε. Πράγματι, αυτή η οικονομία της γνώσης είναι πάρα πολύ σημαντική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις περιφέρειες. Δημιουργεί ε, υψηλή προστιθέμενη αξία και καινοτομία και μέσω αυτών θα πάμε στην ανάπτυξη. Νούμε όμως ότι οι Μητροπόλεις και οι πιο ελκυστικές περιφέρειες είναι αυτές οι οποίες είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να εκμεταλλευτούν όλες αυτές τις δυνατότητες. Θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν ε, τι άποψη έχετε και τι προβλέπετε ώστε οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να μπορέσουν και αυτές ε, να πάρουν το τρένο αυτής της νέας οικονομίας της γνώσης και να μην ε, υστερούν σε σχέση με αυτή την ε, τόσο σημαντική πρόκληση. Τέλος, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, που επισημάνατε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η οποία θα γίνει στη διάρκεια της Προεδρίας σας ε, για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Πρόκειται για μια ανακοίνωση την οποία ε, περιμένουμε, είναι πολύ σημαντική. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ των εξόχως αποκεντρωμένων περιοχών και περιμένουμε από πλευρά σας ισχυρή, σαφή, επιβεβαιωμένη στήριξη υπέρ αυτών των απομακρυσμένων υπερπόντιων περιοχών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βάνο, από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, με, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που παρουσιάσατε τις προτεραιότητες σας ως Προεδρία και είσαστε στη διάθεση Επιτροπής για ερωτήσεις. Ε, εγώ ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε κυρίως όσον αφορά την ε, ιδιαίτερα μεγάλη σημασία της ε, πολιτικής ε, συνοχής και επισημάνατε και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ανάκαμψη μετά την οικονομική κρίση. Από το έκτο πρόγραμμα συνοχής γνωρίζουμε ότι σε ορισμένα κρατημέλη, σε κάποιες περιφέρειες ήταν ακριβώς τα ταμεία τα κονδύλια του Ταμείου συνοχή που βοήθησαν στο να υπάρξουν επενδύσεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, εμείς θέλουμε να υπάρχει μια καλά εξοπλισμένη πολιτική συνοχής για να αμβλύνονται οι διαφορέ στην Ευρώπη ανάμεσα στις περιφέρειες. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις που έχουν τεθεί επιτάπητο για θέματα τέτοια. Παραδείγματο χάρη, το, ο μελλοντικό όγκο ε, τη ε, πολιτική συνοχή και το πολιτέ σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Εσεί θα έχετε τη δυνατότητα να επηρεάσετε τη συζήτηση για το πολιτέ σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό το αναφέρετε στο πρόγραμμά σα εργασία και νομίζω ο συνάδελφο ο το έχει πει ότι μα ανησυχεί ιδιαίτερα ε, το ότι τα πρακτικά της ε, τελευταίας άτυπης συνάντησης ε, των Υπουργών στη Μάλτα. Εκεί ε, αναφέρεται ένα σενάριο ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η πολιτική συνοχής και τα τέσσερα από πέντε σενάρια λένε ακριβώς το αντίθετο. Με ενδιαφέρει λοιπόν να μας πείτε πώς ακριβώς αξιολογείται της ε, πλειοψηφής στο Συμβούλιο, αλλά και τι θα γίνει τελικά με το χρόνο σχεδιασμού. Δηλαδή θα παραμείνουν τα 7 χρόνια φάση προγραμματισμού ή θα γίνει προσαρμογή σε 5 ή 5 και 5 τουλάχιστον ε, όσον αφορά ε, στον πολιτικό κύκλο. Κι άλλο ένα ερώτημα αφορά στο Omnibus ε, για τον οποίο θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη οι τριμερείς διαπραγματεύσεις. Εμείς ε, είμαστε αρνητικοί στο να αφαιρεθούν ε, κονδύλια από την πολιτική συνοχής και να διοχετευτούν το πρόγραμμα ΕΦΣΗ των στρατηγικών επενδύσεων, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το ταμείο ε, έχει τελείως διαφορετικού στόχους από την ε, συνοχή. Και έχουν πραγματικά απεριόριστους πόρους. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω την άποψή σας, γιατί μας ενδιαφέρει η θέση στο Συμβούλιο. Και να ε, πω και εγώ κάτι για το θεματικό, το αστικό θεματολόγιο. Ε, τον Νοέμβρη θα έχουμε το Cities Forum και θα ήθελα να γνωρίζω ε, αν προβλέπετε πότε ε, θα έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για αυτό το αστικό θεματολόγιο Urban Agenda. Δεμάτα. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό για την παρουσία του. Κύριε Υπουργέ, ε, πρέπει να πω ότι στις 27 σελίδες ε, την πολιτική συνεχίστη την αναφέρεται κανένα δυο φορές στη σελίδα 10. Πρέπει να πω ότι είδαμε προγραμματικές δηλώσεις αντίστοιχες και από άλλες προεδρίες, επομένως δεν θα θέλαμε να στιγματίσουμε την Εστονία, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να υπενθυμίσουμε ότι το εξάμεινο που μόλις ξεκινά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πολιτική συνοχή μετά το 2020. Όσον αφορά το θέμα της απάτης, ε, χαίρομαι που αναλάβατε την ευθύνη ε, να ολοκληρώσετε τις ε, διαδικασίες για το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι είναι διεθνή ο χαρακτήρας ε, των παράνομων δραστηριοτήτων που πλήττουν και τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και τις δραστηριότητες τη Ευρωπαϊκής Ένωση συνολικά. Επίσης, όπως αναγνωρίζεται στο έγγραφο, στο δεύτερο ήμιση του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, δημοσιεύσει κάποιες ενδιάμεσες εκθέσεις ε, για τα αποτελέσματα πολύ μεγάλων προγραμμάτων χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων και το Ταμείο Συνοχής και την ε, Κοινή Γεωργική Πολιτική. Και θα αποφασίσει αν θα πρέπει να προτείνει τις δέσμε μέτρο στο πρώτο ήμιση του 2018 ή στο δεύτερο εξάμεινο. Το πρώτο το προτείνει το Κοινοβούλιο και το άλλο δυστυχώ λόγω των καθυστερήσεων φαίνεται ότι θα έχουμε. Αυτά φαίνονται ότι έχουμε από του επιτρόπους Έτιγκερ και Κρέτσου την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, θα ήθελα η Εστονική Προεδρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι εύκολο βέβαια να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση μετά το Brexit, ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ σύντομα τις διαπραγματεύσεις για να γίνει μια κατάλληλη συζήτηση για το νέο πλαίσιο πριν από το τέλος ε, της ε, ε, προεδρία σας. Σας εύχομαι καλή δουλειά παρόλα αυτά. Ευχαριστώ. Έχω κάποιους ακόμα που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τις ερωτήσεις. Ε, η κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Ε, εχθές ε, συναντήθηκα με ε, την μόνιμη αντιπροσωπεία της προομάδας σας που ασχολείται με το Brexit και μίλησα και ε, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και είπατε ότι και είδα ότι αναφερθήκατε και ε, στο θέμα της απλούστευσης και στο θέμα της πρόσβασης της πιστώσης. Είναι κάτι το οποίο το συζητούμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελπίζω να το δούμε στην πράξη, ελπίζω κάποτε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με το Brexit, δεδομένη της δικής σας εμπειρία, ε, η Εσθονία, όπω και η Ιρλανδία είναι μια μικρή χώρα και έχει επωφεληθεί από την ενωσιακή χρηματοδότηση. Εμείς στη Βόρεια Ιρλανδία είχαμε 3,5 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση, είμαστε καθαροί ε, δικαιούχοι. Το Brexit όμως δημιουργεί μια τεράστια απειλή και ένα τεράστιο κίνδυνο στην ε, πρόσφατη πρόοδο που έχει σημειωθεί στο βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας και πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα έχετε να ασχοληθείτε με ζητήματα ε, τέτοια. Ε, η Προεδρία σας δεν είναι τόσο μεγάλη χρονικά όσο και ως άλλες Προεδρίες λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Ο Μισελ Μπαρνιέ άλλοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις ε, με την Βρετανική κυβέρνηση για το Brexit. Το ερώτημά μας λοιπόν είναι το εξή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος που ε, το Κοινοβούλιο και το Προξενείο έχουν συζητήσει αυτό το θέμα ε, για να διατηρηθεί η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής σε ολόκληρο το τμήμα της, να μην έχουμε σκληρά σύνορα στην Ιρλανδία και δεδομένου του ρόλου που έχει παίξει η πολιτική συνοχή για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία και είναι ένα από τα λίγα, ε, ή αν όχι το μοναδικό μέρος το οποίο έχει λάβει τέτοιου είδους ε, ε, χρηματοδότηση υπέρ της ειρήνης. Ε, ήταν τεράστια η πρόοδος, έχουμε καταφέρει την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να υποστούν τεράστια ζημιά ως αποτέλεσμα του Brexit. Θα έχουμε ζητήσει ένα ιδιαίτερο καθεστώς ώστε η Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, ελπίζουμε να υπάρξει μια λύση για την Ιρλανδία από το πρόβλημα του Brexit ελπίζουμε πάση περιπτώσει να παραμείνουμε ε, στη συζήτηση που έγινε υπέρ της διατήρησης ε, της ολότητας της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής ε, ως προς τη χρηματοδότηση και ως τις δυνατότητες που έδωσαν στην ειρηνευτική διαδικασία και στην πολιτική διαδικασία της Βόρειας Ιρλανδίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόπε, τελευταίος ομιλητής. Ačiū ministrė, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, συγχαίρω τον συνάδελφο από την Εστονία για την ανάληψη της Προεδρίας. Μας παρουσιάσετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα Προεδρίας, το οποίο ε, παρουσιάζει και διάφορες εκφάνσεις της ενωσιακής ζωής. Θέλω να πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό θα το εφαρμόσουμε από κοινού. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι η πολιτική συνοχή ε, μόλις τώρα αρχίζει να εφαρμόζεται τόσο στη δική μου τη χώρα όσο και σε άλλες χώρες. Όσοι παίρνουν χρηματοδότηση και εφαρμόζουν προγράμματα ανησυχούν για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής. Στο Κοινοβούλιο είχαμε σχετικές ε, συζητήσεις ε, και σήμερα συζητήσαμε για το θέμα αυτό και τώρα εσείς αναλαμβάνετε την Προεδρία και πάρα πολλά εξαρτώνται από το πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε όλο αυτό το θέμα. Και από εκεί θα εξαρτηθεί και το ποια θα είναι η εικόνα της Ευρώπης το κατά πόσο δηλαδή οι πολίτες ε, των φτωχότερων κρατών θα μετακινούνται προς τα πιο πλούσια κράτη και τα, ή αντίστροφα κατά ε, ε, μέσα σε ίδια τα κράτη οι πολίτες θα μετακινούνται από μικρά χωριά σε μεγάλες πόλεις. Όλα λοιπόν εξαρτώνται από το ποια θα είναι η πολιτική συνοχή και πώς θα εξελιχθεί η περιφερειακή πολιτική. Ίδια δικαιώματα για όλους, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σλόγγαν, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξηγήσετε λιγάκι περισσότερο ε, πώς ακριβώς θέλετε να φέρετε κοντά στους πολίτες ε, την πολιτική συνοχής. Και αυτό μάλιστα σε κάποια κράτη-μέλη όπου δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένη η διάσταση της περιφέρειας. Ε, ξέρετε, κάποιες περιφέρειες χρηματοδοτούνται πάρα πολύ από την Ένωση και άλλες πιο αδύναμες περιφέρειες δεν είναι σε θέση να προσελκύσουν κονδύλια. Και θέλω να σας ερωτήσω, εσείς τι πιστεύετε, πώς πρέπει να κατανέμονται τα κονδύλια συνοχής έτσι ώστε να μην ανακατανέμονται απλά μέσα σε μια χώρα και ορισμένες περιφέρειες να μην υποφελούνται καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Στις ερωτήσεις αυτές ε, ουσιαστικά έχουμε όλο το φάσμα των ε, θεμάτων που απασχολεί και ενδιαφέρει και τους ε, βουλευτές και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ εφαρμόστηκαν όλα τα θέματα τα οποία θα έπρεπε ε, να συζητηθούν ε, τα επόμενα εξάμεινο. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει ένα όμως νήμα το οποίο διατρέχει όλες αυτές τις ερωτήσεις των συντονιστών. Με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να εμπλέξουμε και τους ευρωβουλευτές ε, στις συζητήσεις της Εστονικής Προεδρίας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Με ποιο τρόπο ε, θα διαρθρωθεί αυτή η συζήτηση, πότε θα ξεκινήσει ε, και ήδη σας είπα ότι υπάρχει προγραμματισμένη μία συζήτηση στην ομάδα διευθυντών, σε δύο ομάδες διευθυντών μάλλον, θα γίνουν θεματικές συζητήσεις η κυρία Βέστφαλτ αναφέρθηκε και σε μία έκθεση την οποία ε, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μελετήσουμε ε, το περιεχόμενο και ε, ε, ό,τι μπορούμε να συμπεριλάβουμε θα το συμπεριλάβουμε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα συζητήσει το Νοέμβριο το θέμα της συνοχής. Είναι αλήθεια ότι το χρονοδιάγραμμα είναι λίγο προβληματικό ε, και το γνωρίζετε όλοι σας. Ε, υποτίθεται ότι η 7η έκδοση για τη συνοχή θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο. Τι σημαίνει αυτό. Ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα πρέπει να ξεκινήσουν να συζητώνται ήδη από το Σεπτέμβριο. Αλλά ακόμα δεν ε, ε, είναι έτοιμη η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο αυτή η διαδικασία ε, και η συζήτηση μαζί με το, την έκθεση για την 7η, πολι... Ε, ε, την έκθεση συγγνώμη, για την πολιτική συνοχή και η συζήτηση για τη συνοχή θα γίνει ε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Τι θα κάνουμε στο μεταξύ. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες από πλευρά μα να δούμε αν μπορούν να ενταχθούν στο όλο θέμα τη συνοχή. Ε, πώς θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε και το κοινοβούλιο στις εργασίες μας. Ε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, εξετάζουμε διάφορα ενδεχόμενα, ε, μπορεί να είναι σε επίπεδο συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας, σε επίπεδο διευθυντών, συνεδριάσεις με τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν ε, μπορούμε ε, να ε, αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή. Τώρα, τι σημασία προσδίδουμε στην πολιτική συνοχή εμείς. τεράστια σημασία τα θέματα τα οποία εκκρεμούν όσον αφορά την επόμενη ε, περίοδο και το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε, την πιθανότητα μείωσης του προϋπολογισμού λόγω Brexit, ε, όλα αυτά σαφώς και θα επηρεάσουν ε, τον καθορισμό των εργασιών για τα επόμενα χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε προτάσεις ε, για το πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην επόμενη πολιτική συνεχή ε, και φυσικά εδώ υπάρχουν και ε, τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια που γνωρίζουμε. Τώρα, ο κανονισμός Omnibus, ο τριμερής διάλογος για την πολιτική συνοχή στα πλαίσια του Omnibus θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Ήδη έχουμε προετοιμάσει τις συνεδριάσεις για τον τριμερή διάλογο και ε, ελπίζουμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τόσο πολύ ώστε από 1η πρώτης του 2018 να ξεκινήσει ήδη να εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για την παρούσα ε, προγραμματική περίοδο αλλά και για τη μελλοντική απλοποίηση. Το είπατε ήδη εσείς ότι υπάρχει ομάδα υψηλού επίπεδου που έκανε εξαιρετική δουλειά δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα και σίγουρα οι συζητήσεις ε, που θα γίνουν στις ομάδες εργασίας ε, θα ε, λάβουν υπόψη τους το αποτέλεσμα αυτό. Σας διαβεβαιώ ότι και εγώ θα συζητήσω με τον Σιμ Κάλλας, ο οποίος είναι και πρώην Πρωθυπουργός της Εστονίας και πρώην Επίτροπος και τον γνωρίζετε κι εσείς. άλλα θέματα τώρα τα οποία παρουσιάστηκαν. Έγιναν πολλές ερωτήσεις για το κατά πόσον η πολιτική συνοχής ε, ε, υποστηρίζει όλες τις περιφέρειες ε, και ή μόνο κάποιες πιο ευάλωτες. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Πρέπει να δούμε και τα μακροοικονομικά ζητήματα. Τίθεται διαφορετικά ερωτήματα για τα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή απάντηση. Πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά, να τα μελετήσουμε. Ε, έτσι, εκ πρώτης όψεως μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν υπάρχει καν η απαιτούμενη συνένεση. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό. Άλλωστε υπάρχουν πάρα πολύ περίπλοκα θέματα, για παράδειγμα οι μακροοικονομικές συνθήκες ε, και νομίζω ότι ε, ούτε καν εδώ στην αίθουσα δεν πρέπει να υπάρχει συνένεση για το θέμα. Πρέπει να τα συζητήσουμε λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια απόπειρα να τα δούμε όλοι από το ίδιο κοινό πρίσμα ε, και να δούμε τι θα κάνουμε. Υπήρξαν αρκετά θέματα τώρα που ε, αστική ανάπτυξη, για παράδειγμα. Και αυτό μας απασχολεί. Σίγουρα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, θα υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο ενημερωτικό, αν δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Θα δούμε και τι θα πρέπει να γίνει, αλλά δεν ξέρω αν ακόμα αν αυτό το σημείο θα είναι ενημερωτικό ή αν θα είναι πιο ουσιαστικό. Ψηφιοποίηση τώρα. Αυτό το αγαπημένο μας θέμα είναι τα δικά μας αυτά. Είναι μία από τις προτεραιότητες ε, και ε, εντός της πολιτικής συνοχής. Ε, θα μπορούσα να σας μιλήσω και για μία δράση η οποία εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στην Εστονία ε, και αφορά και τις αιτήσει χρηματοδότησης αλλά και ε, την εξέλιξη της διαδικασίας και την εξέλιξη των προγραμμάτων, την παρακολούθηση των διαδικασιών και ε, την παρουσίαση των συμπερασμάτων. Όλα αυτά τα έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει χαρτί πουθενά. Υπάρχει μία ψηφιακή ταυτότητα η οποία στην Εστονία μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τα πάντα σε επίπεδο εθνικών οργανισμών. Ε, υπάρχει ηλεκτρονική υπογραφή, γίνεται διαχείριση χρησιμεύει για να έχει κάποιο πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω διαδικτύου, ε, σε μία σειρά εφαρμογές ε, κινητών τηλεφώνων και φυσικά μπορούμε να έρθουμε σε επαφή ε, με κυβερνητικές οργανώσεις, οποιοδήποτε πρόγραμμα ή έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή. Και όταν αναφέρομαι στην έξυπνη εξειδίκευση, ε, θεωρώ ότι ενώ στην Ευρώπη δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε κάποιες ηλεκτρονικές λύσεις μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, Εάν δεν μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πολύ δύσκολο θα μπορέσουμε να περάσουμε στα επόμενα στάδια της καινοτομίας. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν στο οποίο θέλουμε να έχουμε κάποια πρόοδο και Ο άνθρωπο μα ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο επίτροπο ε, Άντριου Σάνσιπ, ο οποίο είναι υπεύθυνο για τα ψηφιακά θέματα και είναι ένα πάρα πολύ ικανό άνθρωπο, ελπίζω ότι θα δώσει και αυτό στην κατάλληλη ε, όθηση. Όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο, εδώ μπορώ να σα απαντήσω κάποια πράγματα για ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή και τη χρηματοδότηση. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να επισημάνω ότι η θέση μα είναι προκαταρκτική, προσωρινή. Πιστεύουμε όμω ότι θα ε, καταλήξουμε και στην οριστική μας θέση που δεν θα απέχει και πολύ. Ε, δεν θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να λάβει αναλογικά λιγότερα κονδύλια από ό,τι έχει λάβει μέχρι τώρα. Θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ε, το σημείο αυτό και στη συζήτηση για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όσον αφορά τη πιθανά σενάρια που παρουσιάζονται στη Λευκή Βίβλο, εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος. Εξακολουθώ να φρονώ ότι στα διάφορα έγγραφα ε, προσυζήτηση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πολιτική συνοχή αναφέρεται σαφέστατα και θεωρείται σημαντική. Ε, πιστεύω λοιπόν ε, και ελπίζω πραγματικά ότι αυτή η αρνητική υπόθεση δεν θα υλοποιηθεί. το ελπίζω. Άλλωστε, η Εστονική Προεδρία ε, θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην πάθει τίποτα κακό η πολιτική συνοχή. Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν το Brexit, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω. Αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσει είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω εάν ε, εδώ σήμερα θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Εγώ ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις ε, δεν θα φτάσουν σε ένα σημείο ε, που να ε, βγουν ζημιωμένοι οι πολίτες είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του Ηνωμένου Βασιλείου, είτε της ε, Ιρλανδίας, είτε της Βόρειας Ιρλανδίας. Εμάς το συμφέρον μας είναι να διατηρήσουμε την ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα μπορούμε να συνεχίσουμε να προχωρούμε με επικοδομητικό τρόπο στα θέματα αυτά. Να μην ε, υπάρξει κάποια απομάκρυνση, να μην ξεφύγουμε από το στόχο και να προσπαθήσουμε να τα πετύχουμε όλα αυτά. Τώρα, η έξυπνη εξειδίκευση. Ε, και σε αυτό το θέμα ε, θα υπάρξει ε, μια ανακοίνωση. Η κυρία Μιχαήλοβα νόμιζε ότι θα γίνει την, την επόμενη εβδομάδα. Κάποιοι πίστευαν ότι θα παρουσιαστεί και σήμερα. Δεν ξέρω, αλλά σύντομα τέλος πάντων θα τα καταφέρουμε. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να συζητούμε το θέμα αυτό στην Προεδρία. Εάν ε, ξέχασα κάτι, μπορείτε να μου το ξαναθέσετε και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Θα ήθελα εκ μέρου ε, των μελών ε, της... Διακόπτη Πρόεδρος, ο κύριος Νίστελρο έχετε μία παρατήρηση. Είναι εδώ συνάδελφος, με τον συνάδελφο συζητούσαμε. Από ό,τι κατάλαβα, η Προεδρία θα ενσωματώσει ότι θα λάβουμε ε, πρόσκληση εμείς ως Κοινοβούλιο. Ε, το Ταλίν είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μιλήσατε για τη συναντήση για τις μιλήσατε για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, μιλήσατε για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής και τη σχετική έκθεση. Δεν είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο να μην ε, παραστήσει όλες αυτές τις συζητήσεις. Από ό,τι κατάλαβα θα μας στείλετε μία πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση αυτή. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε κύριε Υπουργέ. Ναι, Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εχθές συναντήθηκα με, κάποιες, με κάποιους συναδέλφους και κατάλαβα από πολλές ε, παρεμβάσεις ότι ε, οι ευρωβουλευτές θα επιθυμούσαν μία πρόσκληση γιατί θεωρούν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θέλουν να συμμετέχουν στις συζητήσεις και θέλουν να εισακουστούν οι απόψεις τους. Νομίζω ότι όταν μιλούμε για την 7η έκθεση πολιτικής συνοχής, δεν μπορούμε να έχουμε επίσημα συμπεράσματα μέχρι ε, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Ε, αυτή τη στιγμή δημοσιευθεί και εφόσον θα έχει γίνει συζήτηση στο Συμβούλιο είναι πιθανό να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Προεδρίας ε, να γίνει μία συνάντηση μαζί σας. Δεν το έχω πει σε κανέναν αυτό, ούτε καν στην Πρόεδρό σας, αλλά είναι πιθανό να έρθω σε επαφή με την Επιτροπή σας και να συζητήσουμε όλες αυτές τις προτάσεις. Αυτή είναι μία από τις δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα είμαστε σε επαφή με την Εστονική Προεδρία θα έχουμε πολλές ευκαιρίες λόγω των τριμερών διαλόγων και όλων των υπολείπων ε, καθηκόντων μας. Θα είμαστε ε, σε στενή ε, αλληλογραφία και επαφή και με τον Υπουργό και με ολόκληρη την Προεδρία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, για τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε για τον ανοιχτό τρόπο με τον οποίο συζητήσατε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι δεν ε, είχατε πει πιο πριν και τα μοιραστήκατε με την Επιτροπή μας. Ε, σας ευχόμαστε, ευχόμαστε μια καλή ε, συνεργασία μαζί σας και με την Προεδρία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Συνεχίζουμε με την κανονική μας ημερήσια διάταξη. Το επόμενο σημείο είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη γνωμοδότηση την οποία, ε, την οποία προετοιμάζει ο κύριος Χέτμαν για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Δεν θα, δεν θα επαναλάβω ολόκληρη την, ε, ολόκληρη την ιστορία, το λόγο του ε, κυρίου Γιούνκερ. Ε, ελπίζω ότι ο εισηγητής μας θα μας παρουσιάσει όλα αυτά τα στοιχεία. Συγγνώμη που υπάρχει θόρυβο στην αίθουσα. Θα, θα, θα σταματήσει πιστεύω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. która spotyka się z zainteresowaniem i jestem przekonany, że pozwoli zmobilizować planowane 100 tysięcy młodych osób do... Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, να έχουμε περίπου 100.000 άτομα και αυτό νομίζω ε, από μόνο του έχει μεγάλη αξία. Άκουσα με ε, μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος ε, Γιούνκα και θέλω να σας πω ότι θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ε, κατόρθωσε να σχηματίσει αυτό το σώμα και να συμμετέχουν ήδη οι πρώτοι εθελοντές. Ακόμα και εάν τυπικά ε, αυτό έχει σχέση με άλλα προγράμματα. Έχουμε λοιπόν ε, μία διαδικασία χωρίς ε, προηγούμενο. Έχουμε μία νομοθετική πρωτοβουλία που δημιουργεί ένα νομοθετικό πλαίσιο. Ε, το σχέδιο είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι κανείς δεν έχει αμφιβολία για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτό το σώμα για την ε, κοινωνία, αυτό το σώμα αλληλεγγύης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός ο εθελοντισμός και χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με βάση τα προγράμματα τα οποία έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ε, θα, μπορούσε να είναι, θα είναι καλύτερο και θα μπορέσουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στην αλληλεγγύη. Ε, θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετίζεται και με το πρόγραμμα Interreg διατηρείται βέβαια η αυτονομία και η ιδιαιτερότητα αυτών των προγραμμάτων. Και θέλω να πω ότι το σώμα της αλληλεγγύης δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα εθελοντισμού, αλλά ε, έχει σχέση και με την απασχόληση, που όμως και αυτή πάλι σχετίζεται με την αλληλεγγύη. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πρόγραμμα και οφείλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όσοι σχετίζονται με το πρόγραμμα ε, δεν ε, θέλουν να αντικαταστήσουν ε, άλλους και δεν θα αντικαταστήσουν άλλους που έχουν ήδη προσληφθεί. Πρέπει να έχουμε κατά νου κάποια σωστή αναλογία. Το δεύτερο που θέλω να πω και έχει σχέση με το σώμα αλληλεγγύης είναι ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για, για την πρώτη απασχόληση ή για τα στάζ. Η, ο εθελοντισμός κατά 80% ε, θα ο θα πρέπει να είναι το 80% και το 20% να είναι κανονική απασχόληση. Το θέμα των ε, στάζ θα πρέπει να αναφέρεται περισσότερο στο έγγραφο. Επίσης, θα ήθελα να ε, αναφερθώ και σε κάποιες ε, τροπολογίες στην πρόταση Επιτροπής. Υπάρχει το περιφερειακό στοιχείο του κανονισμού και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους αδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες και πιστεύω ότι τέλος θα κατορθώσουμε να ε, συντάξουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Ο κατάλογος ε, των σκιωδών εισηγητών δεν μπορώ να πω ότι είναι γεμάτος. Εάν λοιπόν υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Τάκουλα. Ε, στα δικά μου τα χαρτιά λέει ότι εγώ είμαι ο σκιώδης ηγητής. και θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ. Προφανώς τα ε, φινλανδικά δεν είναι μια εύκολη γλώσσα, αλλά επειδή εγώ μιλάω φιλανδικά, θα μιλήσω φιλανδικά. Αλληλεγγύη και συνοχή είναι δύο βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόταση δημιουργεί νομική βάση για το σώμα αλληλεγγύης και προσφέρει την ευκαιρία σε νέους να συμμετέχουν Η συμμετοχή μπορεί να είναι εθελοντική, ε, μπορεί να συμμετέχουν ε, σε αυτό το σώμα με τη μορφή απασχόλησης. Πάντως ε, η συμμετοχή είναι σημαντική. Και πέρα από αυτό, νομίζω ότι υπάρχει και επίσημη ε, επαγγελματική εκπαίδευση. Τίθενται και κάποια ερωτήματα τα οποία δεν ε, ε, ε, διευκρίνησε η συγγήτρια. Ίσως θα μπορούσε να μας τα διευκρινίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, υπάρχει το θέμα της ε, νομικής πράξης. Τι ακριβώς θα επιλέξετε. Θα υπάρχουν συνέπειες, για παράδειγμα, για τη χρηματοδότηση του Εράσμου ΣΥΝ, θα αντανακλάτε με κάποιο τρόπο στο νέο πολυδές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, δεν θα γίνει αυτό ένα αποθεματικό εργαζομένων δευτέρας κατηγορίας, ελπίζω. Ε, με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να το συνδέσετε αυτό με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Ε, τι σχέση έχουν μεταξύ τους, θα παραμείνει η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Ε, θα υπάρχει κάποια ευκαιρία για τους εθελοντές ή ε, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα σημαίνει ότι ε, καταργείται η, ε, ε, το ευρωπαϊκό εθελοντική, η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει επίσης να ξέρουμε και τι ακριβώς σημαίνει εθελοντισμός επισήμως θα υπάρχουν ε, στατιστικά στοιχεία, τι στοιχεία θα καταγράφονται από τους νέους αυτούς, ε, ε, θα λαμβάνουμε υπόψη την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους, τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο για την κινητοποίηση αυτών των νέων. Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις οι οποίες προκύπτουν έτσι εν θερμό, περιμένουμε και κάποιες απαντήσεις, σίγουρα για κάποιες από αυτές έχετε απαντήσεις, αλλά θέλαμε να τις θέσουμε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε από εκεί και πέρα να ε, έχουμε μια γνωμοδότηση ποιότητας η οποία θα απαντήσει σε όλα αυτά τα ε, ε κρεμή ερωτήματα, σε, όλους αυτού, σε όλες αυτές τις παζοκεφαλιές ε, και αυτά είχα να πω λοιπόν ως και ο για την γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χέτμαν για την ε, για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Ζητώ συγγνώμη, η συνάδελφος και η συγγήτρια δεν είναι εδώ και θα την εκπροσωπήσω εγώ. Έχω κάποια, ένα σημείωμα από πλευρά τη. Ε, οι πράσινοι θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι μια ευκαιρία για τους νέους να αποκτήσουν εμπειρία ε, στον εθελοντισμό και να ξεκινήσουν τα δικά τους ε, project. Ελπίζουμε όμως φρέσκο χρήμα να υπάρξει. Αναρωτιόμαστε από πού θα προέλθει όμω. Θα ήταν καταστροφικό λάθος το να πάρουμε χρήματα από πολύ καλά λειτουργώντα προγράμματα όπως το Erasmus Plus ή το ERF. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να παρέχουν φρέσκα κονδύλια για ε, αυτό ε, το ε, σώμα. Εμείς ζητάμε ε, συνύπαρξη με την Ευρωπαϊκή Θελοντική Υπηρεσία χωρίς να διακυβεύεται η ύπαρξή της. Δεν θέλουμε αλληλοεπικαλύψη με υπάρχοντα προγράμματα. Είναι μεγάλη ανησυχία ότι το Σώμα Αλληλεγγύης δεν κάνει τη διάκριση μεταξύ την ε, εθελοντική, μεταξύ της εθελοντικής και της επαγγελματικής του διάστασης. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων και η εθελοντική υπηρεσία δεν μπορεί να το πετύχει αυτό από μόνη της. Χρειαζόμαστε προγράμματα για την τοπική ε, κοινωνία, χρειαζόμαστε προγράμματα ειδικότερα για τους μειονεκτούντες και θέλουμε επίσης το Ευρωπαϊκό ε, Σώμα Αλληλεγγύης να είναι ε, προσπελάσιμο σε όλους και όχι μόνο ε, στους προνομιούχους. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν και πολλές φυσικές καταστροφές που έλαβαν χώρα την περασμένη χρονιά. Έχει ψηλή συμβολική αξία ε, γενικά μια τέτοια πρωτοβουλία. Ε, Περιμένοντα λοιπόν τη γνωμοδέτηση του συναδέλφου που θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο. Εγώ θα κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Με βάση αυτά που είπε ο κύριος Γιούνκερ στη συζήτησή του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016, είπε και παραθέτω, αυτός ο στόχος του σώματος είναι οι νέοι να μπορούν να συμμετέχουν σε αλληλέγγυες πράξεις που αφορούν σε δύσκολες καταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συμμετοχή δεν θα αφορά μόνο τους νέους, αλλά θα συμβάλλει και στις προσπάθειες των τοπικών αρχών και εθνικών αρχών και των ΜΚΟ για να αντιμετωπιστούν διάφορες προκλήσεις και η κρίση. Ε, το πνεύμα της ε, πρωτοβουλίας δεν με βρίσκει σύμφωνη, αλλά παρόλα αυτά συμφωνώ με κάποια από τα στοιχεία που ε, ενέταξε το Κοινοβούλιο στην, στο ψήφισμα του Απριλίου συγκεκριμένα. Δηλαδή εκεί που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στον εθελοντισμό και σε στάζ έτσι ώστε να υπάρχει σαφή διαχωρισμός και εκεί που επίσης αναφέρεται ότι θα πρέπει να ενασχοληθεί το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το εργασιακό περιβάλλον κυρίως όσον αφορά στους ε, εθελοντές ε, ή στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα και κυρίως εκεί που έχω ανησυχήσει είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συστήσει ε, σε μία πρώτη φάση αυτό το σώμα συμπεριλαμβάνοντας ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες και προγράμματα, κυρίως εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα όπως είναι το Erasmus Plus, η Ευρώπη των πολιτών, ε, ο Οργανισμός για τους Νέους, ε, όλα αυτά μπορεί να τα κάνει χωρίς να δίνει άλλη μία ξεκάθαρη άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει σε επίπεδο ανθρώπινο και κοινωνικό. Μία πρωτοβουλία η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη απαιτεί να υπάρχει ε, σαφής ε, εικόνα του, της αλλά και του προϋπολισμού του σώματος αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάλκοβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος ε, που συζητούμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ε, η αλληλεγγύη φέρνει στο νου κάτι το θετικό, κάτι το ευχάριστο. Οι ευρωβουλευτές ε, που εργάζονται στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι πεπισμένοι ότι η αλληλεγγύη είναι ο κινητήρας που θα ε, προωθήσει ε, την ανάπτυξη και θα τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των περιφερειών. Έχω κάποιες ερωτήσεις όμως και θα υποβάλουμε και τροπολογίες ε, σχετικά. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να έχει ένα σύνολο κανόνων, σαφών κανόνων, διαφορετικά θα είναι αμφίσιμο αυτό το έγγραφο. Η ανησυχία μου είναι η εξής. Γιατί μόνο οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, θα είναι σπουδαστές, θα είναι νέοι, ε, νέοι που έχουν ήδη εργαστεί ε, ή θα υπάρξει κάποιο όριο ηλικίας. Αν υπάρχουν και άλλοι που ενδιαφέρονται για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, μπορούν εκείνοι να προσπαθήσουν ε, να έχουν πρόσβαση και να ρωτιέμαι τι είδους δραστηριότητες θα υπάρξουν. Θα είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ε, θα είναι ε, ε, απασχόληση, πώς ακριβώς θα, θα έχουν τα πράγματα και θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις, τα ερωτήματά μου αυτά. Θα θέλαμε πάντως να υποστηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μισλέ. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Μιχέλης εμείς ε, πιστεύουμε γενικά ότι αυτό το πρόγραμμα ε, το να υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον ε, διότι αντιμετωπίζει σωστά το πρόβλημα. Βέβαια, για μας υπάρχουν κάποια σημαντικά ερωτήματα και πρέπει να σας πω το εξής. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα καλά κατά πόσον αυτό το σώμα θα διαφοροποιείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού. Από ό,τι φαίνεται σε αυτό το πρόγραμμα ε, το βάρος δεν αποδίδεται στον εθελοντισμό. Δίδεται σημασία σε στάζ, σε θέσεις απασχόλησης για τους νέους και πρέπει να σας πω, δεν είμαι πεπισμένη για το κατά πόσον ε, ε, αυτό είναι και το πιο λογικό εντάξει δεν μπορεί κανείς ε, να διαφωνεί με το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καλώνει να εφαρμόζει τέτοιου είδου προγράμματα. Από την άλλη βέβαια δεν έχω καταλάβει ακριβώς ε, στο ποιος θα κάνει τελικά τη διαφοροποίηση το τι είναι ένα πρόγραμμα αλληλεγγύης και τι είναι μια προσφορά για δοκιμαστική άσκηση, για στάζ όπως λέγονται. Και τίθε για μένα το εξή ερώτημα. Μία θέση απασχόλησης. Γιατί ε, στην περίπτωση αυτή περιορίζεται σε 12 μήνες και στην πρωτοβουλία του κυρίου Γιούγκερ αυτό που ενδιαφέρει είναι να προσφέρονται στους νέους σταθερές θέσεις απασχόλησης και ε, πολύ συχνά τίθεται το θέμα των, ε, της χρηματοδότησης και εδώ όμως από ό,τι φαίνεται ε, υπάρχουν οκτώ προγράμματα που ήδη τρέχουν και εμείς ως πράσινοι ενδιαφερόμαστε να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα γίνει τελικά η χρηματοδότηση. Ο κύριος Βανίστελρο παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι πάντοτε ενδιαφέρον είναι στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιφερικής Ανάπτυξης να προβληματιζόμαστε επί τέτοιων πρωτοβουλειών και να προσπαθήσουμε να πάμε ακόμη παραπέρα στο πλαίσιο αυτής της νέας δραστηριότητας. Γιατί στην Ευρώπη διαπιστώνουμε ότι Πρέπει να τονιστεί η συμμετοχή των ε, πολιτών ε, περισσότερο, ε, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα και κοινωνικής φύσεως και περιβαλλοντικές καταστροφές και θεομηνίες και πρέπει να μπορούν να διαδραματίζουν ένα ρόλο πιο ενεργό. Το θέμα είναι σε ποιον απευθύνεται τέτοιου είδους δραστηριότητα και πώς θα τα καταστήσουμε όλα αυτά πιο συγκεκριμένα γιατί δεν δίνουμε τη δυνατότητα στις ε, περιφέρειες, στις πόλεις, ε, στους κατοίκους ε, να αναλάβουν τα ενία αυτής πρωτοβουλίας και να τους δώσουν την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και εμείς να είμαστε απλώς ένας διάβλος επικοινωνίας, γιατί έχουμε την τάση να το ξεχνούμε οι άνθρωποι αυτοί είναι έτοιμοι να ε, συμμετάσχουν, είναι έτοιμοι να πούν την άποψή τους, ε, είναι μία εμπειρία και τέτοιου είδους δραστηριότητα θα έπρεπε να συνεισφέρει και στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των ε, πολιτών της. Ο καθένας πρέπει να αισθάνεται ότι είναι σε θέση να συμμετέχει και νομίζω ότι αυτό υπερβαίνει την απλή συμμετοχή. Πρόκειται για μία εμπειρία και στο πλαίσιο της Επιτροπής μας Νομίζω ότι θα έπρεπε και εμείς να δεσμευθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Για ποιο λόγο η ε, επιτροπή, υπάρχει και η επιτροπή των περιφερειών, υπάρχει η επαφή μας με τους επιτρόπους, ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θα μπορούσαμε να επιμείνουμε στην προώθηση τέτοιου είδους πρωτοβουλειών και να ε, δούμε πώς οι άνθρωποι θα μπορούσαν να συμμετέχουν μέσω βιντεοδιάσκεψης. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό σώμα σημαίνει ότι θέλω να συμμετέχουν σε μια νέα πρωτοβουλία. Ε, ίσως στο παρελθόν να το έχουμε ξαναπροσπαθήσει και να μην υπήρξε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Επιτροπή μας όμως πρέπει ε, να τονίσει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν την συλλογική οικειοποίηση αυτού του, του πνεύματος της πρωτοβουλίας. Ε, μιλάω για το κοινό, μιλάω για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ίσως θα έπρεπε να ακολουθήσουμε ένα νέο μοντέλο, γιατί αν ακολουθούμε συνέχεια τις ίδιες μεθόδους, στο ίδιο αποτέλεσμα θα καταλήξουμε. Νομίζω λοιπόν ε, ε, θέλουμε να αφήσουμε τα άστρα να λάμπουν. Ε, πρέπει όμως να το καταφέρουμε αυτό. Αξίζει τον κόπο. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαλνίστερλόι. Έχουμε τώρα εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ από δύο γενικές διευθύνσεις. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Δεν ε, έχει κάποιος διάθεση να ξεκινήσει. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ρόμπερτ Φράνσερ εγώ Είμαι στη Γενική Διεύθυνση Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και είμαστε υπεύθυνοι για τη σύσταση ε, του σταδίου της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος Ελληνικής. Θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις ε, ε, που ετέθησαν. Ε, κάποια πράγματα είναι προφανή γιατί μας θέτουν συχνά τέτοιες ερωτήσεις. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ιδέα ε, αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματος Ελεγγύης και το γεγονός ότι αναπτύξατε αυτή την ευκαιρία ε, να μπορέσουν οι νέοι να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς την αλληλεγγύη και στη συμμετοχή τους ε, στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Τώρα στις ερωτήσεις. Υπήρξε μια ερώτηση από αρκετά μέλη του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ε, συνέπειες ε, και την επιρροή του προγράμματος Erasmus ε, Συν και πώς επηρεάζεται από το σώμα αλληλεγγύης. Ξέρετε ότι για πάνω από 20 χρόνια υπάρχει Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ουσιαστικά μεταφέρουμε τις δραστηριότητες ε, οι οποίες αναπτύχθηκαν εντός του πεδίου εφαρμογής ε, για τη ε, ε, εθελοντική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και μεταφέρονται και τα κονδύλια. Αυτό φαίνεται και στην νομοθετική πρόταση, αλλά δεν κάνουμε απλώς μεταφορά των κονδυλίων και αλλαγή στην ονομασία. Προσθέτουμε και την επαγγελματική διάσταση, δηλαδή τη μαθητεία και τις θέσεις εργασίας, αλλά προσφέρουμε και νέες μορφές εθελοντισμού και προστίθεται και δυνατότητα όχι μόνο δραστηριότητες σε άλλη χώρα, αλλά και εντό της χώρας. Πρέπει να σας πω ότι τίναμε δίκονους ε, στα όσα μας έλεγε το κοινού στη δημόσια διαβούλευση πριν κάνουμε την πρόταση και ήταν σαφές ότι έπρεπε να φροντίσουμε δύο πτυχές κατά την εφαρμογή. Την ποιότητα να μην περιορίσουμε δηλαδή την ποιότητα των θέσεων εθελοντισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, ε, αντίθετα να τα βελτιώσουμε, να προσέξουμε την ποιότητα της μαθητείας και των θέσεων εργασίας που προσφέρουμε και να υπάρχει και σαφής διάκριση μεταξύ τους. Και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε. Ταυτόχρονα ε, προσέξαμε ιδιαίτερα ώστε να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να μην αποκλείει κάποιους. Έχουμε λοιπόν συμπεριλάβει και κάποιες νέες μορφές δραστηριοτήτων, πιο βραχυπρόθεσμες, που επιτρέπουν λοιπόν σε νέους ανθρώπους να προσφέρουν ε, θελοντική εργασία για σύντομο χρονικό διάστημα, να γίνονται ομαδικά, ε, να συμμετέχουν δηλαδή συλλογικά ε, νέοι άνθρωποι ιδίω από πιο ε, ευάλωτο παρελθόν περιβάλλον νιώθουν καλύτερα να συμμετέχουν συλλογικά κάποιου ε, και επίσης να μην είναι μόνο μονοπλήρους απασχόλησης, αλλά ε, να μπορούν και στο χρόνο τους να προσφέρουν. Νέοι άνθρωποι λοιπόν στείνουν κάτι σε τοπικό επίπεδο για να προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία στον ελεύθερο χρόνο τους. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι ε, ένα επιπλέον έναυσμα πέραν των οικονομικών κινήτρων για τη συμμετοχή και των ευκαιριών. Υπάρχει και η δυνατότητα να μην αποκλείσουμε κανέναν από το πρόγραμμα. Τώρα, οι εφαρμοστικές δομές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι οι ίδιες εκτελεστικές δομές που έχουμε και στο Erasmus Sin. Άρα η εφαρμογή δεν γίνεται απευθεία εδώ ε, στις Βρυξέλλες μέσω των εκτελεστικών υπηρεσιών μας, αλλά κυρίως μέσω ενός συστήματος εθνικών υπηρεσιών που ε, βρίσκεται στα κράτη-μέλη. Και αυτό μας εξασφαλίζει μια πολύ ε, στενή παρακολούθηση ε, τα, για τα μικρής κλίμακας ε, έργα τα οποία είχαμε και στο προηγούμενο πρόγραμμα Erasmus η Οι εθνικές υπηρεσίες, για να έρθω εδώ στις ερωτήσεις του ποιος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, θα είναι αρμόδιες για όλο το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Θα καλύψουμε λοιπόν και την πτυχή, την επαγγελματική και τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 33.000 ε, εγγεγραμμένους ε, στην ιστοσελίδα που έχουν εκφράσει την ε, προθυμία τους να συμμετέχουν σε θελοντικές δραστηριότητες ή σε κάποιες θέσεις εργασίας. Ε, παρεπιπτόντως, όταν εκφράζουν ε, την επιθυμία τους για το σε ποιες δραστηριότητε θέλουν να συμμετέχουν, το 86% λέει ότι θέλουν να συμμετέχουν είτε στο ένα είτε στο άλλο. Επομένως, τους ενδιαφέρουν και οι δύο διαστάσεις, που είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, διότι δείχνει ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κάτι και για να ε, εκφράσουν αλληλεγγύη τους. Ε, βεβαίως αυτή η καταχώρηση των νέων ανθρώπων που θα αποτελέσουν και το βασικό σώμα αυτού του σώματος ελληνική μας δίνουν και τη δυνατότητα να συνεργαστούμε μαζί τους όχι μόνο όταν ε, θα ε, πάνε στο χώρο της δραστηριότητας, αλλά και πριν και να τους υποστηρίξουμε και μετά. Διότι ο στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν στη δράση της δραστηριότητες, για να τους βοηθήσουμε, για παράδειγμα, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αργότερα. Ε, για τον προϋπολογισμό. Αναφέρθηκα ήδη στις δραστηριότητες ε, που αφορούν ε, τον εθελοντισμό. Αυτές έχουν συμπεριληφθεί ε, και μεταφερθεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Έχουμε και τα σχετικά κονδύλια, 198 91,1 εκατομμύρια. Έχουμε κάποιο προπολογισμό ακόμα στο Erasmus για δραστηριότητες εθελοντισμού οι οποίες δεν εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Επομένως και τα δύο προγράμματα θα έχουν ακόμα ε, δραστηριότητες εθελοντισμού και θα υπάρχει υποστήριξη και για αυτές. Και επειδή ακριβώ θα είναι οι ίδιοι οι φορεί αυτοί που θα εφαρμόσουν και τι δύο δραστηριότητε, πιστεύουμε και θα θέλαμε ε, να έχουμε τις ίδιες διαδικασίες και τον ίδιο εξοπλισμό, να μην υπάρχει ε, χαμηλής τιμής, εθελοντισμός, ε, ε χαμηλής αξίας και δαπανηρός από την άλλη. Θέλουμε να έχουμε μία ομαλή προσέγγιση και για τις δύο πλευρές και για τους οργανισμούς. Κάποιος αναφέρθηκε στη σημασία της τοπικής κοινότητας και το πώς μπορούν να βοηθήσουν οι νέοι άνθρωποι και τη σχέση με τα όσα κάνουν και τα όσα γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η φιλοδοξία μας. Αν ε, δείτε, μία από τις αλλαγές που έχουμε στους γενικότερους στόχους του προγράμματος είναι ότι δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στους νέους ανθρώπους και όχι μόνο στις οργανώσεις, αλλά και στις ανάγκες των ε, κοινοτήτων. Ήδη λοιπόν από τώρα προσπαθούμε να ε, συνδέσουμε τις δραστηριότητες των νέων με τα όσα συμβαίνουν στον περίγυρό τους και θα θέλαμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στο θέμα αυτό. Ένα από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται συχνά και οδηγούν σε σύγχυση είναι η σύνδεση του πρώτου σταδίου που έχουμε στο 2017 ε, που βασίζεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο και βασίζεται σε αυτά τα 8 προγράμματα τα οποία κινητοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα της ελληνικής. Πρέπει να σας πω ότι το 2017 εφαρμόζουμε ακόμα 8 διαφορετικά προγράμματα τα οποία ε, ήδη ε, συμβάλλουν σε αυτή την ιδέα αλλά δεν πάβουν να είναι 8 ξεχωριστά προγράμματα που το σημείο σύνδεσης είναι αυτό ο αριθμός των νέων ανθρώπων που έχουν καταχωριστεί και θέλουν ε, να συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τον προπολογισμό αυτών των προγραμμάτων και έχει προβλεφθεί και έχει συμφωνηθεί ε, ε, στους αντίστοιχους φορείς διακυβέρνησης αυτών των προγραμμάτων. Υπήρχε επίσης και μια ερώτηση για το γιατί επικεντρωνόμαστε μόνο στους νέους ανθρώπους και ποιος είναι ο ορισμός των νέων ανθρώπων. Χρησιμοποιούμε τον ορισμό ε, για άτομα ηλικίας 18-30 ετών και ε, ε, επικεντρωνόμαστε μόνο στους νέους γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η γενιά στην οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Είναι ευάλωτη, ε, σε κάποιες περιπτώσεις τους έχει πλήξει η οικονομική κρίση με πιο σοβαρό τρόπο και μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των αναγκών της κοινωνίας ε, και να μην ε, χάσουν το στόχο τους. Υπήρχε και μια ερώτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα τι δραστηριότητες θα πρέπει να κάνουν Δίπλα στην πρόταση για τον κανονισμό έχουμε και μια, ένα έγγραφο εργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο εξηγούμε λίγο πιο αναλυτικά τι δραστηριότητες ε, και πώς ε, θα πρέπει να διατυπώνονται. Υπήρχε και μια ερώτηση γιατί η μέγιστη διάρκεια είναι μόνο 12 μήνες και γιατί δεν έχουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο λόγος είναι για να μην θεωρηθεί αυτό ως ένα μέσο της αγοράς εργασίας που υποκαθεστά θέσεις εργασίας ή ότι είναι μια ενεργός πολιτική αντιμετώπισης της ανεργίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαφορετικά μέσα για αυτό το θέμα και αντιστοίχως έχουν και τα κράτη-μέλη. Εμείς λοιπόν εδώ ασχολούμαστε μόνο σε ε, θέσεις εργασίας και μαθητείας, σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλληλεγγύη. Εάν ε, μελετήσετε διεξοδικά την πρόταση, τον έφερε και ο πρώτος ομιλητής, ε, τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την επαγγελματική διάσταση είναι πολύ χαμηλότερα από τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για την εθελοντική διάσταση, γιατί θεωρούμε ότι ο εθελοντισμός είναι ε, ένας από τους ε, καλύτερους τρόπους έκφρασης αλληλεγγύης, το ισχυρότερο μέσο για να εκφράσει κανείς την αλληλεγγύη του υπήρχε και το ερώτημα της οικονομικής σταθερότητας. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε μια ξεχωριστή νομική βάση. Με αυτή την πρόταση Προσφέρουμε ασφάλεια δικαίου και σταθερότητα για τα μέσα τα οποία αναφέρονται εδώ, για τα 351 ε, εκατομμύρια 500.000 για τα πρώτα τρία χρόνια για να δραστηριοποιηθούν αυτοί οι οργανισμοί σε θέματα αλληλεγγύης και ε, να προβλέψουν και ε, πόσες ευκαιρίες θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και για την ιδέα να συμπεριτέχουν οι πόλεις και οι περιφέρειες. Αυτό ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε, διότι με τη δημιουργία αυτής της ομάδας των ε, νέων ανθρώπων που έχουν κίνητρα ενεργαστών, δεν θα έχουμε απλώ ε, ένα σύνολο ανθρώπων για να επιλέξουμε, αλλά ε, θα είναι και αυτοί οι οποίοι θα διαδώσουν το μήνυμα για την αλληλεγγύη, για την Ευρώπη και έτσι θα έχουμε περισσότερη συνοχή στην κοινωνία μα. Πρόκειται για πάρα πολύ καλή ιδέα και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και μαζί σα ε, για το θέμα αυτό στο μέλλον. Ελπίζω να μπόρεσα να διευκρινίσω τα περισσότερα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ λεπτομερής εξήγηση. Κυρία Ρίτλερ, μήπως θέλετε και εσείς να πάρετε το λόγο, να προσθέσετε κάτι. Um, no, uh, my colleague. Η συνάδελφος... Ε, ο συνάδελφο, συγγνώμη, Ρομπέρτο, ήδη έγραψε την κατάσταση πολύ καλά. Κάτι ακόμη ίσω θα μπορούσα να προσθέσω. Καταρχά, ε, εγώ είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και θα ήθελα μία ακόμη φορά να τονίσω ότι η επαγγελματική διάσταση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν, είναι, δεν έχει ως κύριο στόχο να αντιμετωπίσει την ανεργία μεταξύ των νέων. Έχουμε άλλου είδους μέσα για να το κάνουμε αυτό. Έχει μια πολύ ευρύτερη ένα πολύ ευρύτερο ε, πεδίο ε, ε, εφαρμογής της υποστήριξης απασχόλησης των νέων, 20.000 θέσεις απασχόλησης και θέσεις άσκησης δεν είναι αρκετές για να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Είναι απλώς μια επιπλέον δυνατότητα για τους νέους ε, να λάβουν ε, ε, ποιοτικές ευκαιρίες απασχόλησης συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Ένα ερώτημα υπήρχε επίσης και για το φθηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό είναι και για μας μια πολύ σοβαρή ανησυχία. Πρέπει η τοποθετήσεις να είναι ε, ποιοτικές, ε, Ζητούμε όλες οι περίοδοι μαθητείας ε, να συνάδουν με το πλαίσιο για την μαθητεία, το οποίο το έχουμε ήδη αναπτύξει και επίση θέλουμε να είναι αμοιβόμενες, αμοιβόμενες από τον εργοδότη και για την απασχόληση θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να συνάδουν με τους εθνικούς κανονισμούς ε, έναν ελάχιστο, ένα βασικό μισθό ε, όταν ε, ισχύει κάτι τέτοιο βέβαια. Επίσης προγραμματίζουμε εταίρους της αγοράς εργασίας αλλά και δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας θέλουμε να συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στην όλη διαδικασία γιατί υπάρχει ψηλό επίπεδο ευφυΐας ε, στο πλαίσιο της, ε, ε, του εργατικού δυναμικού και μετά την τοποθέτηση των νέων μπορούμε μακροπρόθεσμα να τους εντάξουμε στην αγορά εργασίας και με άλλες δραστηριότητες, όπως ε, για παράδειγμα αντιστήχηση των νέων με τις κατάλληλες θέσεις απασχόλησης ε, και αμαθητίας. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Χέτμαν, έχετε το λόγο για να ε, συνοψίσετε τη συζήτηση. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Ε, τέτσαν κάποιες ερωτήσεις, δεν απαντήθηκαν όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ προφανώς ε, δεν είμαι ε, εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε άλλο, έχω αρκετές επιφυλάξεις όσον αφορά στο έγγραφο που εξετάζουμε. Αλλά πρέπει να πω ότι το έγγραφο αυτό συντάχθηκε σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα και είναι ένα ποιοτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι πρέπει να συγχαρούμε εκείνους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εργάστηκαν επί του εγγράφου. Ο αξιότιμος κύριος Τάκουλα έκανε μία ερώτηση σχετικά με το μέλλον μετά το 2020. Αυτό όμως δεν αφορά το έγγραφο, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα έγγραφο που αφορά την περίοδο 2018-2020 και έχουμε να κάνουμε και με ένα έγγραφο ε, το οποίο απαριθμεί τους, ε, τις οικονομικές, ε, τους οικονομικούς πόρους για το ΕΡΑΣΜΟΣΥΝ. έχει σχέση και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με το πρόγραμμα Live, όπως επίσης και με το Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη. Ως εκ τούτου όλα αυτά ε, αναφέρονται μέχρι το 2020 με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Το τι θα γίνει μετά το 2020 θα το συζητήσουμε αργότερα, εν το χρόνο. Κατόπιν, το τι θα γίνει ε, σε σχέση με, το, ε, με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Από την ε, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία θα πάρουμε όλες αυτές τις ε, δραστηριότητες που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ υπάρχει και ο εθελοντισμός που έχει σχέση με τρίτες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου εδώ υπάρχει απόλυτη συμπληρωματικότητα των δράσεων. Η κυρία Σμόλκοβα. έθεσε μία ερώτηση που αφορά στους τομείς ε, στους οποίους θα αναπτυχθεί αυτός ο εθελοντισμός ε, αφορά και στις ε, δοκιμαστικές ε, περιόδους. Ε, όλα αυτά έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, με τις ε, φυσικές καταστροφές, με την υγεία, την δημιουργικότητα, τον πολιτισμό, την φυσική, σωματική αγωγή, κοινωνική, παροχή κοινωνικής βοήθειας. Όλα αυτά αναφέρονται με απόλυτες, με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αλλά και αυτά βέβαια μπορούμε να τα συζητήσουμε αν θέλουμε να διευρύνουμε το πλαίσιο. Και όπως σας είπα, έχουμε αυτό το νέο εργαλείο, το οποίο ε, δεν θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί κανείς ε, για το εργατικό δυναμικό. Το σήμα ποιότητας των ε, οργανώσεων που θα καλύψουν αυτές τις θέσεις απασχόλησης αλλά και την δοκιμαστική εργασία. Αυτό ε, κατά την άποψή μου είναι μια εγγύηση για να αποφύγουμε καταστάσεις όπου θα μπορούσαν να προκύψουν ε, καταχρήσεις και θα μπορούμε λοιπόν να εγγυηθούμε ότι αυτοί οι νέοι ε, θα μπορέσουν πραγματικά να εξελιχθούν. Κατόπιν, ποιος θα μπορεί να συμμετέχει. Ε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μας είπε ότι θα μπορούν να συμμετέχουν άτομα μέχρι τις ηλικίες των 30 ετών, αλλά έχουμε και την περίπτωση των ε, νέων σε μειονεκτική θέση. Αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο ε, αυτού του νέου σώματος είναι άτομα με αναπηρία ή με δυσκολίες στη μάθηση ή προβλήματα υγείας και αυτά περιγράφονται με πολλές λεπτομέρειες. Κατά την άποψή μου λοιπόν ε, όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και για να ολοκληρώσω. Κατανοώ ε, την, ε, τα επιχειρήματα όσον αφορά στην ισορροπία ανάμεσα στο 80% και το 20% υπέρ βεβαίως του εθελοντισμού και είμαι απόλυτα σύμφωνος ότι αυτό το εργαλείο δεν μπορεί να εξαλείψει την ε, νεανική, την απασχόληση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή την ηλικιακή ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ πιστεύω ότι ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος θα βρει μία θέση απασχόλησης με βάση αυτό το πρόγραμμα, ήδη αυτό είναι προσθέμενη αξία. Το να υπάρχει σταθερή θέση απασχόλησης για ένα νέο είναι κάτι τελείως διαφορετικό από, την, από τον απλό εθελοντισμό. Πολύ ωραία, θα τα ξαναπούμε μετά τις ε, θερινές διακοπές. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση και πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι η γνωμοδότηση που έχει προετοιμάσει ο συγητής μας, ο κύριος Βαλκαρσέλ Σίσο, σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης. Παρακαλώ κύριε Σίσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το είπα και σήμερα το πρωί, αλλά επιτρέψτε μου να το επαναλάβω και σήμερα το απόγευμα. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιτρέψατε να ε, μεταφέρουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία κανονικά έπρεπε να έχει γίνει σήμερα το πρωί, αλλά για λόγους που σας εξήγησα δεν, μπορούσε να, δεν μπορούσα να είμαι εδώ νωρίτερα. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν, ε, ειλικρινά. Η γνωμοδότηση αυτή τονίζει τη σημασία που έχει η πολιτική συνοχής ως μέσο το οποίο είναι σε θέση να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης ε, και ε, συνεισφέρει την ανάπτυξη των περιφερειών και των πόλεων μας και είναι και ένα μέσο το οποίο ε, υποβοηθά τις επενδύσεις. Ε, θεωρώ ότι πάντα είναι κατάλληλη στιγμή για να τονίσουμε τη σημασία της προόδου στην οικονομική και κοινωνική συνοχή ε, και να γεφυρώσουμε χάσματα μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών. Σήμερα όμως είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ αυτό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει δύσκολες στιγμές και δεν σας λέω βέβαια και τίποτα που δεν γνωρίζετε, αλλά είναι αλήθεια ότι η πολιτική συνοχή είναι ο βασικός τρόπος που έχουμε για να δώσουμε όθηση στην ανταγωνιστικότητα και να υλοποιήσουμε την αλληλεγγύη που είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει να αμβλύνουμε τις ανισότητες που δημιούργησε η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να σας πω ότι το κείμενο ε, καλύπτει αρκετές πτυχές κλειδί, όπως για παράδειγμα την ανάγκη ε, να συνεχίσουμε να εξετάζουμε πώς θα μπορέσουμε να διαβιβάσουμε τα αποτελέσματα ε, της πολιτικής συνοχής ε, στους πολίτες. Πρέπει επίσης να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε όθηση στην αστική διάσταση των ευρωπαϊκών περιφερειών, χωρίς όμως να αφήσουμε πίσω την διάσταση της υπαίθρου. Επίσης, λέμε ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και τις πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες καινοτομία και έρευνας, ιδίω εκείνες οι οποίες ε, αφορούν τους νέους. Τέλος, ε, κάτι εξίσου σημαντικό με τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτό το έγγραφο να χρησιμοποιηθεί για να συνεχίσει να προωθεί την πολιτική συνοχή. Και όλα αυτά για να έχουμε μια αποτελεσματική κότερη χρήση των πόρων, όπως για παράδειγμα πρωτοβουλίες ε, για την ε, απασχόληση των νέων, που πραγματικά θα βοηθήσουν ε, για την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι νέοι δεν είναι απλώς το μέλλον της Ευρώπης, εγώ θεωρώ ότι είναι το παρόν, διότι αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεών μας. Για να ολοκληρώσω, το έγγραφο αυτό τονίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η πολιτική συνοχή να διαθέτει πιο ευέλικτους μηχανισμούς, καθώς επίσης και να ε, προωθήσει και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Ε, Συνολικά η γνωμοδότηση που σας παρουσιάζω σήμερα το απόγευμα τονίζει πόσο σημαντική είναι η συνοχή για να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα είναι εύρωστο, έξυπνο, βιώσιμο ε, και θα, δεν θα αποκλεί κανέναν και δεν θα αφήνει πίσω κανέναν και να αφορά όλες τις περιφέρειες διότι ε, στην πραγματικότητα αυτό είναι ο στόχος όλων των οικονομικών πολιτικών που διέπουν την Ευρωζώνη. Αυτά λοιπόν ε, ήθελα να πω, αυτή είναι η παρέμβασή μου και αυτή η γνωμοδότηση ε, αυτά περιλαμβάνει και τώρα από εδώ και πέρα θα ακούσω με ιδιαίτερη προσοχή τις παρεμβάσεις σας, οι οποίες σίγουρα θα χρησιμεύσουν για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε το αρχικό κείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Να δώσω το λόγο στους Σκιώδης, η κυρία Μπρέσο. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο για αυτή, αυτό το πρώτο σχέδιο. Νομίζω ότι Υπάρχουν πάρα πολλά ε, πολύ ενδιαφέροντα θέματα σε αυτήν την ε, έκθεση και θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια θέματα και μετά θα δούμε πώς θα μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε σε τροπολογίες. μπορούμε να δούμε τους προϋπολογισμούς ε, της ε, ζώνης του ευρώ. Και ίσως θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, περισσότερο στη σημασία που έχει η πολιτική συνοχή για τη ζώνη του ευρώ. Και σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο η Ευρωζώνη τουλάχιστον όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, το υπάρχει ένα κοινό έχει ανάγκη που να αποφεύγουν τις ανισορροπίες. Και εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η πολιτική συνοχή για όλες τις περιοχές μπορεί να βοηθήσει στο να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις στην ίδια τη ζώνη και να σταθεροποιηθεί το ευρώ. Είναι σαφές ότι αυτή η προοπτική είναι καθοριστική σημασία και η πολιτική συνοχή ε, καλύπτει όλες τις ε, ζώνες Όλε όλες τις περιοχές της Ευρωζώνης. Ακόμα και εκεί που υπήρξαν ε, μεγάλα σοκ. Η Ευρωζώνη χρειάζεται ε, την ανατροπή της κατάστασης πρέπει να περάσουμε σε μια ταχεία διαδρομή ε, σταθεροποίησης και για να επιτευχθεί η σταθεροποίηση είναι καθοριστική σημασία να προβλέπουμε έναν ικανοποιητικό προπολογισμό στη ζώνη του ευρώ έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινητροδοτήσουμε ε, την ε, σύγκληση να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ε, κρατών μελών, να προσπαθούμε να επιφέρουμε σταθερότητα σε ολόκληρη τη ζώνη. Ε, ο ισολογισμός της ζώνης του ευρώ μπορεί να επηρεάσει και την ικανότητα των κρατών να απορροφήσουν ασύμετρα και συμμετρικά σοκ. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η πολιτική της συνοχής από μόνη της δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό την πολιτική συνοχή, στην πολιτική συνοχή δεν μπορεί κανείς να φορτώσει την ε, έξοδο από την κρίση, γιατί η πολιτική συνοχή έχει ως στόχο να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα κάποιων περιοχών. Άρα δηλαδή ο στόχος είναι μικροοικονομικός, μικροοικονομική παρέμβαση όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ε, Άρα δηλαδή είναι μια πολιτική η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι μικροοικονομική παρέμβαση και αφορά μεμονωμένους τομείς. Ενώ οι παρεμβάσεις για εξωτερικά σοκ, όπως είναι μια μεγάλη κρίση, αυτή είναι ξεκάθαρα μια μακροοικονομική παρέμβαση. Εμείς πρέπει να πούμε ότι η πολιτική συνοχή μπορεί να επιτύχει συγκεκριμένα πράγματα εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ. Ο προϋπολογισμός της ζώνης του ευρώ μπορεί να επιτύχει άλλα πράγματα τα οποία θα παρεμποδίζουν την απόκληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή και την απόκληση ανάμεσα σε συγκεκριμένες περιοχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μας πείτε εσείς την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των τροπολογιών. Είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε κάποιο τρόπο να συμφωνήσουμε. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ. Τόμασιτς παρακαλώ. κυρία Τόμασιτς, έχετε το λόγο. Έχουμε προγράμματα τα οποία πρέπει να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα. Δυστυχώς όμως έχουμε το, την κληρονομιά της κρίσης ε, που είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για την ε, ανάπτυξη. Η επιτυχία των πολιτικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση εξαρτάται επίσης από τους μηχανισμούς ε, στρατηγικού σχεδιασμού και χρηματοδότησης των ε, προγραμμάτων. Βεβαίως, ε, σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά εξαρτώνται και από την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι προϋποθέσεις είναι βέβαια η εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών με τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα και η συγκέντρωση σε εκείνα τα προγράμματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν τα κονδύλια θα πρέπει να διοχετεύονται στις πιο αδύναμες περιοχές και όχι σε όλες τις περιοχές. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για τη μακροοικονομική σταθερότητα αλλά και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες ε, είναι προς όφελος της μείωσης ανεργίας. Ευχαριστώ κυρία Νικολάη από τους φιλελεύθερους. Δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να σας παρουσιάσω την άποψή της και την συμβολή της στη συζήτηση. Καταρχάς θα ήθελε να επισημάνει ότι υποστηρίζει τη θέση του εισηγητή και τον ευχαριστεί για την καλή δουλειά του, θα ήθελε να κάνει τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση, η βασική έκθεση δεν καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μόνο τα μέλη της Ευρωζώνης ε, στην μακροοικονομική προσέγγιση, οικονομικές πολιτικές ή γενικές γραμμές καλύπτουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, για παράδειγμα συνθήκη του Μάστριχτ ή το δημοσιονομικό έλλειμμα κλπ. Η έκθεση αναλύει κάποιες πολιτικές Ευρωζώνης, οι οποίες πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις γενικές αρχές ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Από την άποψη της συνοχής, το ζήτημα το οποίο πρέπει να τεθεί είναι το εξή Τι ρόλο η περιφερειακή πολιτική διαδραματίζει για την Ευρωζώνη. Δυστυχώς υπάρχουν απόψεις που θεωρούν ότι η πολιτική αυτή απλώς μειώνει, τις, αμβλύνει τις διαφορές ε, στην ανάπτυξη μεταξύ των παλαιότερων και των νεότερων περιφερειών. Ε, η απάντησή μου, λέει η κυρία Νικολά, είναι ότι η συνοχή είναι ένα καλό εργαλείο για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και πρέπει να διατηρηθεί για όλους όλα αυτά μπορούμε να δεχθούμε την ευελιξία και την ανάγκη απλούστευσης των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Αυτές ήταν οι σκέψεις της κυρίας Νικολάη ως της εισηγήτριας και τώρα θα συνεχίσουμε με την κυρία Μίχελς που είναι η επόμενη σκιώδη εισηγήτρια. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι η έκθεση ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Ε, ο κύριος Σίσο το είπε, κυρίως ε, διότι η πολιτική συνοχή τοποθετείται σε σωστή προοπτική και προβάλλεται ως ένα σημαντικό στοιχείο για την εξορροπημένη εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσθέσω, πρώτον, όλοι μας ε, συμφωνούμε ότι η πολιτική συνοχή ε, πράγματι μπορεί να αμπλύνει τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες κρίσης, αλλά έχει και όρια. Αυτό που δεν μπορεί να επιτύχει είναι να εξαλείψει πλήρως τα λάθη που έχουν γίνει. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να αλλάξει πολιτική, να ξεφύγουμε από την πολιτική της λιτότητας και να περάσουμε σε αναδιάρθρωση χρέους, ε, στην αναδιανομή του πλούτου ε, και μέσα από τα διορθωτικά ταμεία αλλά και άλλα εργαλεία. Επίσης, συμφωνούμε ως προς το ότι η πολιτική της συνοχής ε, προφανώς και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ε, προκλήσεις, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να περιμένουμε από την πολιτική αυτή χωρίς επιπρόσθετα κονδύλια να αναλαμβάνει όλο και περισσότερα καθήκοντα. Σε αυτή τη γνωμοδότηση νομίζω θα πρέπει να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά αυτά τα οποία έχει ήδη πει πολλές φορές η Επιτροπή ε, Περιφερειών, δηλαδή είναι σημαντικό να υπάρχει συνέργεια ανάμεσα σε διάφορα εργαλεία, όμως να μην υπάρχει υφέρπουσα μετάβαση ε, στην πολιτική, της πολιτικής συνοχής ε, σε μια επενδυτική πολιτική η οποία θα προσανατολίθει κυρίως σε ιδιωτικές και κερδοφόρες επενδύσεις. Και τέλος, ε, η ευρύτερη διασύνδεση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και με ε, συστάσεις αναχώρα, αυτό η δική μου πολιτική ομάδα το απορρίπτει. Γιατί και μόνο αυτή η χρονική ε, αλληλουχία των συστάσεων αναχώρα παρεμποδίζει τη λειτουργία της πολιτικής συνοχής και αυτό μας το έχουν επιβεβαιώσει πάρα πολλοί εκπρόσωποι. Εξάλλου, πολλές συστάσεις όπως παραδείγματο χάρη η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης ή ε, απελευθέρωση πολλών τομέων, αυτά αντιβαίνουν στους στόχους της ε, πολιτικής συνοχής. Και ειδικά το δικό μας το Κοινοβούλιο πρόσφατα απέρριψε την μακροοικονομική ερεσιμότητα. Και αυτά τα έκρινα ότι είναι στοιχεία του πολιτικού συντονισμού. Κύριο Σκάρλετς. Push the wrong button. Συγγνώμη, πάτησα λάθο κουμπί. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμεί ε, επικροτούμε ε, την έκθεση και θα κάνουμε και εμεί τι παρατηρήσει μα σχετικά με τη γνωμοδότηση. Καταρχάς, αναφέρεται η ανάπτυξη. Εμείς θα θέλαμε και την ε, αηφόρο ανάπτυξη να τονίζεται περισσότερο στο κείμενο. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό να το προσθέσει κανείς και να βελτιώσει το μήνυμα. Εμείς χαιρετίζουμε τα μέτρα της ε, τρέχουσας προγραμματικής περίοδου για να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η πολιτική με, το, με τη στρατηγική για το 2020 για την ε, ανάπτυξη. Η, ο χρονισμός όμως του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων είναι διαφορετικός γιατί δεν έχουν το ίδιο ε, στόχο. Ίσως θα έπρεπε ένας κύκλος μικρότερος μπορεί να αποδυνάμωνε τις, ε, την επιτυχία των διαρθρωτικών αλλαγών στον, στις περιφέρειες. Μία ακόμη παρατήρηση, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα, ε, η ανάκαμψη, ε, αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο αρνητικό στις περιφέρειες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν υπάρξει αποδυνάμωση πολιτικής συνοχής γιατί είναι η βασική δικαιούχη. Κάτι ακόμη αρνητικός αντίκτυπος των μέτρων την κοινή γνώμη ε, ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης τονίζουμε ότι ο σημαντικός αριθμός ε, χωρών που λαμβάνουν συστάσεις ε, δεν, μπορούν, δεν μπορεί να, εφαρμοστεί χωρίς την έγκριση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρξει ένα σχεδιασμό μια διαδικασία σωστή συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε το ρόλο των πολιτών και των Δήμων στην επένδυση, ε, στο ε, κλίμα, ε, στις προσαρμογές, στην αλλαγή του κλίματος. Βέβαια, εγώ ως, εμείς ως πράσινοι τονίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να συμπεριλάβει την αηφορία στον ευρύτερο κύκλο προγραμματισμού των πολιτικών. Επενθυμίσουμε επίσης ότι η μείωση της ανισότητας, η βελτίωση της ε, πιο περιεκτικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να αυξηθούν, να φτάσουν το 30% των κονδυλίων συνοχής σε κάθε κράτος μέλος και να γίνεται πρικοδότηση τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα ε, κατά το οποίο δεν μειώνεται ο κύκλος πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα την συνεργασία μεταξύ των ταμείων, πρέπει να υπάρχει υπάρξει καλύτερη συνεργασία, όχι μόνο μεταξύ των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και του ορίζοντα 2020, αλλά και την, ε, ε, ε, το Connecting Europe Facility, τα κοινωνικά ταμεία, όπως επίσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Όλα αυτά πρέπει να συμπληρώνουν το ένα το άλλο, όμως δεν θα έπρεπε να μειωθεί η στρατηγική συνοχή, ούτε η μακροπρόθεσμη προοπτική πολιτική της, πολιτικής συνοχής. Και τέλος, αυτό που για μας είναι πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι οι αεροζεόντιες αρχές ε, της πολυεπίπεδης ε, διακυβέρνησης, ε, του να συμπεριληφθεί διάσταση του κλίματος στις πολιτικές, έχουν δείξει τη σημασία τους για την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων και πρέπει η χρήση των κονδυλίων να βελτιωθεί προς αυτή την κατεύθυνση στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο για να σχολιάσει. Κυρία Μαλέτιτς, ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τις ε, παρεμβάσεις τους και τον εισηγητή μας για την γνωμοδότηση. Αυτή η συζήτηση για τις οικονομικές πολιτικές ε, λαμβάνει χώρα και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν είναι εύκολο να κάνουμε τη διάκριση των οικονομικών πολιτικών ε, ε, της Ευρωζώνης και των κρατών μελών εκτός Ευρωζώνης γιατί το μείγμα οικονομικής πολιτικής είναι το ίδιο για κάθε κράτος μέλος, επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση, έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία, ε, ε ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, ε, την ε, ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Ε, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν αποτελούν ένα μείγμα για όλες τις χώρες της Ένωσης και πρέπει να δούμε πώς θα τονίσουμε τον ρόλο της πολιτικής συνοχής, γιατί αυτή η πολιτική είναι πολύ οριζόντια, αφορά όλα αυτά τα θέματα ε, σε ένα σωστό οικονομικό μείγμα που χρειάζεται σε κάθε κράτος μέλος ώστε να μπορέσει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, ε, ε, την ανάπτυξη των θέσεων απασχόλησης, ε, την αύξηση των θέσεων απασχόλησης επίσης. Εμείς θέλουμε ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να τονίσουμε ότι μία ισχυρή Ευρωζώνη είναι μία προϋπόθεση για μία ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε η ισχυρότερη Ευρωζώνη χωρίς όλα τα κρατη και όλες τις περιφέρειες και αυτό είναι ο ρόλος πολιτικής συνοχής, να ενισχύσει όλες τις περιφέρειες ε, προκειμένου να απαλληφθούν αυτές οι ανισότητες και οι διαφορές. Ε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ... Ε, πρέπει να, κάνουμε μια ηχηρή έκκληση για ένα σωστό μείγμα πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γιατί η πολιτική συνοχής δεν αφορά μόνο τις επενδύσεις αλλά και την ε, ε ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Πολύ σύντομα, ε, επειδή έχουν ε, λεχθεί τα περισσότερα, ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Εγώ νομίζω ότι... Αν δει κανεί τι διάφορε αξιολογήσει, θα διαπιστώσει ότι τα τρία τέταρτα των συστάσεων αναχώρα είναι στα χέρια των πόλεων και των περιοχών, των περιφερειών. Έτσι λοιπόν, το να προτείνει κανείς ε, το ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασωθεί η Ευρωζώνη, αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Κατόπιν, ε, δεν υπάρχει ένα έγγραφο ε, σχετικά με τις, τις Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Θα πρέπει τουλάχιστον να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία μορφή του ευρωπαϊκού προεκλογισμού. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να λεχθεί, να είμαστε σαφείς. Ε, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι να πάρουμε ένα κομμάτι της συνοχής και με τρόπο αυτό να δώσουμε κίνητρα στην Ευρωζώνη. Ε, δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική για όλες τις περιφέρειες. Επίσης, η συνοχή είναι στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν είναι πρόγραμμα ούτε εργαλείο. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να κάνει κανείς κάτι λιγότερο σε επίπεδο συνοχής. Αυτό δεν πρέπει να το συγχαίουμε. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το θέμα των περιφημών externalities, των εξωτερικών αθέσεων. Ο συνάδελφός μου έρχεται από τη Βουλγαρία. Οι επενδύσεις ε, στη Βουλγαρία αποφέρουν ε, ωφέλη στις άλλες χώρες. Έχει κατατεθεί ένα έγγραφο από τις χώρες Βίζεγκάρτ ε, στο Συμβούλιο ε, σχετικά με τις εξωτερικές ε, συνθήκες και υπάρχουν εκεί κάποια στοιχεία Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ Συνοχής ακούσαμε πολύ προσεκτικά τον κύριο Μοσκοβισή ε, που είπε ότι η συνοχή σημαίνει ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι χώρες ε, θα έπρεπε να μπορούν να γίνουν μέλη. Αυτά είναι θεωρία νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια. Πάντως σημασία έχει η συνοχή να είναι ένας ξεχωριστός στόχος και προϋπολογισμός. και ίσως θα πρέπει να έχουμε ε, και ένα έγγραφο από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, γιατί δεν ξέρω εκείνοι ε, τι σκοπεύουν να κάνουν. Uh, θα συνεχίσουμε τώρα με παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θέλω να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο κύριος Βανίστελ Ρόι και να του πω ότι έχουμε το σχέδιο της έκθεσης. Λυπάμαι αν δεν το έχετε πάρει, αλλά έχει ε, μοιραστεί. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you very much, Ευχαριστώ πάρα πολύ αξιότιμη κυρία Πρόεδρε και αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να συγχαρεί ε, τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για την γνωμοδότηση αυτή. Λαμβάνουμε γνώση, όπως ε, γνωρίζετε, ε, η χρήση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις οικονομικές πολιτικές Ευρωζώνης αναφέρεται στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 21 Μαΐου 2017 δημοσιεύτηκε η σχετική έκθεση και οι προτάσεις, τα μέτρα που προτείνονται μεταξύ άλλων σκοπό έχουν να ανατρέψουν τις κοινωνικές ε, ανισότητες και διαφορές ε, εντός και μεταξύ των κρατών μελών και κάποια βήματα προτείνονται ένα πακέτο εργαλείων ε, για τη σύγκληση, ε, σταθερότητα, σταθεροποίηση, ε, συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων και έχει προτείνει την επέκταση του ΕΕ για γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει τριμερής διάλογος σχετικά και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αναβιώσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις ε, και παράλληλα γίνεται και επιπλέον δουλειά για να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα με ε, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ένωσης. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη δουλειά σας ε, για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά για να συνοψίσετε τη σημερινή συζήτηση. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον ε, για τη γνωμοδότηση. Έλεγα προηγουμένως ότι θα μπορούσατε κι εσείς ε, με τις παρεμβάσεις σας να συνεισφέρετε και σίγουρα θα εμπλουτίσουμε αυτό το κείμενο να σας πω ότι σίγουρα δεν έκανα λάθος, διότι από αυτά τα οποία άκουσα από εσά βλέπω ότι ε, θα καταφέρουμε να εμπλουτίσουμε το αρχικό κείμενο το οποίο σας παρουσίασε. Ε, αυτό ακριβώς θέλαμε και νομίζω ότι αυτό ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι επετεύχθη. Υπάρχει ένας κοινό παρανομαστής ε, σε όλες τις παρεμβάσεις, ε, αν ε, ήθελα να κάνω και μία σύνοψη, αλλά πάρα πολύ λακωνική. Υπάρχει ο εξή κοινό παρανομαστής, η συνογή. Η συνοχή είναι ισότητα και ισότητα σημαίνει ότι η συνοχή πρέπει να μειώσει τις ανισότητες. Επομένως, δεδομένου ότι υπάρχει συγκεκριμένη ε, πολιτική συνοχής είναι σαφές ότι συνεχίζουμε η επιτυχία θα έρθει αργά ή γρήγορα, αλλά ε, θα ε, έχει σχέση και με την καταπολέμηση της ένδυας. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από ισχυρές περιφέρειες και ε, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη η Ευρωζώνη να διαθέτει μία σειρά από μέσα τα οποία θα μειώσουν αυτές τις ελλείψεις ισορροπίας, ε, θα μειώσουν αυτές τις ταλαντώσεις οι οποίες δημιουργούνται ε, και δημιουργούν διακυμάνσεις μεταξύ περιφερειών που αντιμετώπισαν με μεγαλύτερο τρόπο την κρίση και είδαν να μειώνεται η ανταγωνιστικότητα. Θεωρώ ότι όλα αυτά μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στο κείμενο, ε, γιατί εντάσσονται πλήρως στο κείμενο το οποίο σας παρουσίασα προηγουμένως. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η ισορροπία, όπως επίσης είναι απαραίτητο κατά συνέπεια να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, όχι μόνο στις περιφέρειες αλλά και στα κρατη Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η γνωμοδότηση αυτή να μπορέσει να ε, περιλαμβάνει και πτυχές όπως για παράδειγμα η επίλυση των σφαλμάτων στην οικονομική διάρθρωση των κρατών μελών. Και είναι σαφές ότι η γνωμοδότηση ε, θα δοθεί σε ε, μία έκθεση της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ε, επομένως, ε, μιλάμε εμεί για τη συνοχή, αλλά φαίνεται ότι δεν διευρύνεται ο τίτλος και το περιεχόμενο όσων συζητάμε. Στην πραγματικότητα εμείς δεν ε, επιλέξαμε τον τίτλο. Ο τίτλος είναι της έκθεσης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εμείς απλώς γνωμοδοτούμε επί της εκθέσεως, επομένως δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα στον τίτλο πέραν της αρχικής έκθεσης. Ε, συμφωνώ απόλυτα ε, ότι υπάρχει ανάγκη να διευρύνουμε την έννοια της ανάπτυξης ε, και να προσθέσουμε τον όρο βιώσιμος, βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό θα κάνουμε. Και είναι αλήθεια ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε την ε, οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης ε, με τα όσα θα μπορούσαν να ισχύουν εκτός Ευρωζώνης. Και εδώ έχετε και το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής είναι μια πολιτική ε, η οποία τέμνει κάθετα όλες τις υπόλοιπες πολιτικές. Και φυσικά ε, πρέπει να υπάρχει ενότητα, το έλεγε ο κύριος Βανίστερ ε, πρέπει να υπάρχει ενότητα στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική συνοχής πρέπει να χρηματοδοτεί όλες τις περιφέρειες, διότι η συνοχή, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι απλώς αίτιο και η συνοχή δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Η συνοχή είναι ένας στόχος ή, όπως πολύ σωστά έλεγε ο κύριος Φανίστερ Ρόι, είναι ένας ξεχωριστός στόχος από το σύνολο του προπολογισμού της Ένωσης, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να θεωρείται ως ενιαίος. Είναι λοιπόν ένας στόχος, είναι αυτοσκοπός. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλους εκείνους που ε, προσέφεραν κάποιες νέες ιδέες, οι οποίες σίγουρα θα συμπεριληφθούν σε αυτή τη γνωμοδότηση, διότι αυτό θέλουμε να την εμπλουτίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρκάρλ Λεσίσο. Το τελευταίο το οποίο έχω να σας πω είναι να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για τη γνωμοδότηση αυτή είναι Τετάρτη 19 Ιουλίου 12 το μεσημέρι θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση στις 7 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη λοιπόν, 19 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Αυτά για τη γνωμοδότηση αυτή. Λύεται λοιπόν η συνεδρίαση και θα περάσουμε τώρα στο τμήμα της συνεδρίασης που θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Ε, όσοι δεν συμμετέχουν στην ομάδα των συντονιστών θα πρέπει να αποχωρήσουν και θα συνεχίσουμε με τους συντονιστές.